Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Άρχεται η συνεδρίαση. Οι αρχές αρμόδιες από την Πορτογαλία μου απίθυναν έτοιμα ανάκληση της άρσης ασυλίας του κυρίου Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες στο πλαίσιο ποινική διαδικασίας εις βάρους του από τις ε, αρχές δίωξης της πόλης του Πόρτο. Το σχετικό αίτημα έχει αναπαιμφθεί στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη την κοινή συζήτηση για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Γυναίκες στα Διοικητικά Συμβούλια. και δίνω το λόγο σε μία από τις συντάκτριες, την κυρία Γκαρσία Πέρες. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έλλειψη εκπροσώπησης ε, των γυναικών στα διάφορα πεδία της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής είναι ε, εκδήλωση της ανισότητας στην κοινωνία. Άρα χρειάζεται να προωθήσουμε την πολιτική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. <clears throat> το 2013 το κοινοβούλιο μας έλαβε θέση έναντι της ε, πρότασης της Επιτροπής για την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να υπάρξουν υποχρεωτικές ποσοστώσεις εκπροσώπησης των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο ούτω ώστε και στον οικονομικό τομέα λοιπόν να υπάρξει ίση εκπροσώπηση. Έκτοτε πέρασαν πέντε χρόνια. Πέρασαν διάφορες προεδρίες και το θέμα αυτό έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να προωθήσουν μια πιο ίση Ευρώπη, καταλαβαίνοντας ότι μια Ευρώπη πιο ίση πρέπει οπωσδήποτε να είναι μια Ευρώπη όπου είναι πραγματικότητα ίση εκπροσώπηση των γυναικών σε όλου του τομεί τη οικονομική ζωή. Έπρεπε να αλλάξει η κυβέρνηση στην Ισπανία για να δοθεί μια όθηση και στο Συμβούλιο, ούτω ώστε να επιδιώξουμε επιτέλους να υπάρξει μια συμφωνία για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιούροβα για την όθηση που διαπιστώνω ότι δίνει, ούτω ώστε η Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να επιτρέψουν να ολοκληρωθεί πριν από το τέλο τη ιδίας μια πρωτοβουλία για την ισότητα εκπροσώπηση που είναι θεμελιώδη. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε τα δικαιώματα των γυναικών να συνεχίσουν να καθυστερούν να εφαρμοστούν. Οι γυναίκε πρέπει οπωσδήποτε να εκπροσωπούνται ισότιμα, να υπάρχει ισότητα ευκαιριών. Και το κοινοβούλιο μα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει σαφή θέση και να, να καλέσει την Ρουμανική Προεδρία να κάνει την τελευταία προσπάθεια, ούτω ώστε όπω ε, και η κυβέρνηση τη Ισπανία που προωθεί την ε, πρωτοβουλία αυτή, ούτω ώστε να καταφέρουμε οι γυναίκε να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Είναι θεμελιώδε για να προχωρήσουμε προ μια Ευρώπη πιο ίση και πιο δίκαιη. Σα ευχαριστώ πολύ. Συντάκτη επίση η κυρία Χάουταλα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και είναι πιστεύω πολύ σημαντική η στιγμή τώρα να διαπιστώσουμε πως ουδής λόγος μας αποτρέπει από την υιοθέτηση αυτής της οδηγίας του 2012, από την εισαγωγή αυτής της οδηγίας, που θα επέβαλε την υποχρέωση καταχωρημένες ε, ε, εταιρείες, επιχειρήσεις να φτάσουν στο 40% ποσοστό για τα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Με καταπλήσει το ότι ορισμένα κράτη-μέλη επικαλούνται ακόμη την επικουρικότητα. Πώς το κάνουν αυτό. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις ευρωπαϊκές που δρούν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και πέραν αυτής. Επομένως οπωσδήποτε είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, το αντικείμενο της οδηγίας. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η διαφορά, η συμπερίληψη και η ποικιλία μεταξύ αυτής βέβαια και της διάσταση του φύλου και για την ε, διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των στρατηγικών των επιχειρήσεων. Τρίτον, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν ικανές γυναίκες. Αυτό είναι μια πρόφαση μόνο μιας ε, νοοτροπία στην οποία επικρατούν οι άντρε. Ναι, μπορεί να μην είναι ορατέ οι γυναίκε γιατί μερικέ φορέ δεν έχουν αυτή τη νοοτροπία ή τη συμπεριφορά που ε, προέρχεται από την ε, νοοτροπία όπου επικρατούν την ανδροκρατούμενη, αλλά πάντως είναι εξίσου ικανές με τους άντρες τουλάχιστον για να ανταποκριθούν σε προκλήσεις. Και έτσι πρέπει και σε αυτό το βαθμό να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις. Είχαμε πει αρχικά εθελοντικά, στην εισαγωγή των γυναικών, όπου διαπιστώσαμε στο το 2017-2018 ήταν μόνο το 26% των διοικητικών συμβουλίων γυναίκε τις μεγαλύτερε από τι καταχωρισμένε επιχειρήσει Ευρωπαϊκής Ένωση, μεγάλη διαφορά από το 7,5% στο 43% που αποδεικνύει πως χρειάζονται μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα μας οδηγήσουν στην αναρμόνιστη σημαντική αυτή πτυχή. Ευχαριστώ την Ισπανική κυβέρνηση, η οποία επιτέλους έριξε μια δεύτερη ματιά στην υπόθεση αυτή. Και ελπίζω ότι με την ε, Προεδρία της Ρουμανίας θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την πρόταση και πριν από τις ευρωεκλογέ να μπορέσουμε να διακηρύξουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει ένεργα μια σύγχρονη και επιχειρηματική κουλτούρα και νοοτροπία με ισότιμη ε, προώθηση και ε, εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, γιατί υπάρχει ένας λόγος να μην συμβαίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους Συμβουλίου τώρα η Υφυπουργός κυρία Σότ την οποία και ευχαριστώ για την παρουσίαση της εδώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, μεγάλη χαρά που σας βλέπω εδώ σήμερα για αυτή τη σημαντική συζήτηση. Ξεκινώντας θέλω να πω πώς η ισότητα των φύλων εγγράφεται στο επίκεντρο του οράματος για την Ευρώπη του Συμβουλίου σε πολλές διακήρυξεις του Συμβούλου έχει επιβεβαιώσει αυτή την προσήλωση, αλλά και στην νομοθεσία που αναπτύξαμε σύν το χρόνο από κοινού με το Κοινοβούλιο. Και επίσης θέλω να υπενθυμίσω τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που από κοινού ανεκήρυξαν Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017. Η ισότητα των φύλων λοιπόν έχει μεγάλη σημασία εδώ η ισότητα των φύλων, ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να προάγεται σε κάθε τομέα συμπεριλαμβανομένη και της εκπροσώπησης σε όρους αγοράς εργασίας και τις συνθήκες απασχόλησης και προαγωγής στη σταδιοδρομία. Άνδρες και γυναίκες έχουν δικαίωμα σε ίση αμοιβή για δουλειά ίσης αξίας. Αυτή η προσήλωση βεβαίως και καταχωρίζεται και προέρχεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες αλλά και από τις εθνικές μας νομοθεσίες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε όμως. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο, την τελευταία πεντηκονταετία αλλά και περισσότερο βλέπουμε ότι υπάρχουν πρακτικές των οποίων ακόμη δεν έχουμε τον έλεγχο ή την επιστασία. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω σαν παράδειγμα ότι υπάρχει ακόμα σημαντική διαφορά ως προς την αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, 16,2 ποσοστιαίες μονάδων και πάντα είναι χαμηλότερες οι αμοιβέ των γυναικών από, τους, από αυτές των ανδρών. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί ισότητα. Το ζήτημα λοιπόν της αμοιβή θα το ε, καλύψουμε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου που αναμένουμε να υιοθετηθεί στον Συμβούλιο Άψκο τον Ιούνιο. Για να υλοποιηθούν όμως και οι άλλες ε, υποσχέσεις του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων χρειαζόμαστε δράση από την Επιτροπή, από τους συνομοθέτες, από τα κράτη-μέλη. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα μας ζητήσατε συγκεκριμένα να ε, σχολιάσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία που θα βελτίωνε την ίση εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των ε, επιχειρήσεων. Με λύπη μου σας λέω σήμερα ότι δυστυχώ, όπω άλλως το γνωρίζετε υπάρχει σχετική μειοψηφία στο Συμβούλιο. Η τελευταία μας συνεδρίαση για το θέμα αυτό είχε λάβει χώρα υπό την Προεδρία της Μάλτα το 2017. Η συζήτηση δε δεν συζητήθηκε έκτοτε ε, επισήμως από το Συμβούλιο όπως έχει τώρα η κατάσταση παραμένει δηλαδή σε αδιέξοδο αυτή η υπόθεση πλην όμως ευρεία είναι η συνένεση στην Ευρώπη ως προς την ανάγκη για προαγωγή της ισότιμης εκπροσώπησης των φύλων στα διοικητικά συμβούλια όσο και αν έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα κράτη-μέλη γιατί δεν αμφισβητείται η βάση αυτή της στόχευσης και έτσι η Ρουμανική Προεδρία στοχεύει να διευκολύνει τις συζητήσεις και συνομιλίες επί του Συμβουλίου προκειμένου να διερευνηθούν υπεραιτέρω ε, διάβλη για πρόοδο. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην πρόταση για μία οδηγία για, την, ε, για το συγκερασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου για γονείς ε, και εδώ θα ήθελα να πω ότι η συνομιλίες μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου οδήγησαν σε μια προσωρινή συμφωνία στον έκτο τριμερή διάλογο που έλαβε χώρα στις 24 Ιανουαρίου. Επιτυχία η οποία κατέστη δυνατή και χάρη στην εξαιρετική πρόοδο που ε, οφείλουμε στη Βουλγαρική και Αυστριακή Προεδρία. Η διευκόλυνση λοιπόν του συνδυασμού οικογενειακού και επαγγελματικού βίου είναι τεράστιος πυλώνα τη πολιτική απασχόληση. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνουμε του πολίτε μα να συγκεράσουν τον επαγγελματικό με τον οικογενειακό βίο, πράγμα το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό και λόγω της δημογραφικής κατάστασης και των εξελίξεων στην αγορά εργασίας όμως. Αφενός λοιπόν πρέπει να καταστήσουμε να εξασφαλίσουμε πως η Ευρώπη θα έχει γυναίκες με την υψηλή τους κατάρτιση και τις δεξιότητές τους ικανές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, πράγμα το οποίο έχει και οικονομική σημασία και αντίκτυπο, ταυτόχρονα είναι και τα δικαιώματα και από την άλλη θα πρέπει οι γυναίκες και οι άνδρες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παιδιά χωρίς να πρέπει να κάνουν την επιλογή μεταξύ του να είναι γονείς ή να έχουν μια θέση εργασίας. Και βεβαίως επισημαίνω ότι πολύ πιο συχνά οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τέτοια επιλογή. Έτσι λοιπόν, εάν οι εργαζόμενοι που έχουν οικογένεια έχουν κατάλληλα δικαιώματα για άδεια γονεακοί ή άλλοι και αυτά τα δικαιώματα ε, είναι κατανεμένα τόσο στους άντρες όπως και στις γυναίκες, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο πρέπει και τα εθνικά συστήματα να τροποποιηθούν. Στη γυναίκα, στην Ευρώπη δεν μπορεί να πει κανείς ότι μία λύση μπορεί να ισχύει για, το, κάθε, για όλα τα κράτη αδιακρίτως. Ε, έτσι λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές πραγματικότητες και κοινωνικά συστήματα μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αλλά και να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Αυτές ήταν κάποιες από τις σκέψεις που εκλήθημε να συζητήσουμε κατά τις συνομιλίες για την οδηγία για την εξορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Εύκολη δεν ήταν η συζήτηση, αλλά χαίρομαι ότι, διότι ευρέθη μία λύση η οποία εξασφαλίζει με την α, βελτίωση των ε, απαιτήσεων και των προδιαγραφών τη δυνατότητα για την εξορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και ελπίζουμε και το Κοινοβούλιο είναι ικανοποιημένο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τώρα την το λόγο θα λάβει η Επίτροπος κυρία Γιώργοβα, την οποία και ευχαριστώ για την παρουσία της. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο επειδή έθεσε το σημαντικό αυτό θέμα στην σημερινή ημερήσια διάταξη. Είμαι ευγνώμων για την ε, στήριξή σας στην πρόταση της Κομισιόν που στόχο έχει να βελτιώσει την ισορροπία των δύο φύλων σε εταιρικά διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών. Εδώ και πέντε χρόνια σχεδόν είμαι τώρα Επίτροπος για την ισότητα των φύλων και είμαι υπερήφανη για την συλλογική μας δουλειά, ειδικά για την οριστικοποίηση του πακέτου για την ισορροπία μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού βίου. Ανησυχώ όταν το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα λέει στην ε, τελευταία του έκθεση, στον δείκτη του, ότι σε κάποιους τομείς ε, πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά. Όταν ε, δημοσιεύσαμε τα πιο πρόσφατα νούμερα, δεν έκρυψα την απογοήτευσή μου για τις εξελίξεις αυτές, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουμε. Ο δείκτης ισότητας των φύλων δείχνει πως η ισότητα στην λήψη αποφάσεων εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από όλους τους άλλους τομείς που αξιολογήθηκαν στον δίκτυ παρά την νομοθεσία σε κάποια κράτη που εντωμεταξύ εγκρίθηκε. Όλοι γνωρίζουμε τις μελέτες που δείχνουν σαφώς τα ωφέλη της ποικιλομορφίας ε, στα διοικητικά συμβουλία. Οφέλη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία βεβαίως. Η Κομισιόν βεβαίως ε, παραμένει προσιλωμένη στην οδηγία αυτή. Οι γυναίκες παρά τις ικανότητες τους ε, συνεχίζουν να έχουν να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην ε, είσοδό τους στα διοικητικά συμβουλία και σε ηγετικέ θέσεις. Η οδηγία αυτή θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την πρόσβαση ταλαντούχων γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις και να επιταχύνουμε την οικονομική ανάπτυξη. Όταν αποκτήσουν εξουσία οι γυναίκες ε, θα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο θα διευρύνει την ισότητα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως πρόκειται για μια πρόταση αναλογική και ευέλικτη, φιλική προς την επικουρικότητα που δίνει μεγάλη ευελιξία στα κρατημέλη για το πώς θα επιτευχθεί αυτή η πρόοδος. Επίσης, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο είναι ουδέτερο ως προς τα φύλλα. Αφορά το φύλλο το οποίο εκπροσω... υποεκπροσωπείται ε, όταν έχει ανάλογα προσόντα, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες. Και βεβαίως ε, τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να διατηρήσουν τα υφιστάμενα μέτρα που έχουν για να βελτιώσουν την ισορροπία των φύλων στα ΔΣ. Σύμφωνα με τους αριθμούς μας, τα κράτη τα οποία έχουν περάσει την νομοθεσία σημειώνουν κάποια πρόοδο. Όσα δεν έχουν την νομοθεσία έχουν απλά κολλήσει. Βλέπουμε λοιπόν τον θετικό αντίκτυπο της ε, νομοθεσίας αυτής σε πολλά παραδείγματα. Η πρόταση της ε, Κομισιόν έχει ευρία στήριξη από το Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι και επίσης έχει την στήριξη της ε, πλειοψηφίας των κρατών μελών. Κατά την άποψή μου, μπορούμε να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση και θα επαναλάβω αυτό το οποίο υπόθηκε, ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη από την ε, Ισπανική κυβέρνηση ε, τους οποίους είχα επισκεφθεί ούτως ή άλλως ε, πρόσφατα και αυτό μας δείχνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για να πείσει και τις χώρες εκείνες που ακόμα είναι αντίθετες. Και επίσης ε, βασιζόμαστε ιδιαίτερα και στην Ρουμανική Προεδρία που επίσης είναι πολύ αποφασισμένη. Εν ώψη του Συμβουλίου του Μαρτίου σκοπεύουμε να ξεμπλοκάρουν οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και η υπουργό ανέφερε και το Συμβούλιο του Ιουνίου που πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το επέσχυντο αυτό ζήτημα του μισθολογικού χάσματος. Οπότε η Κομισιόν ελπίζει ότι η Ρουμανική Προεδρία θα καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για το θέμα αυτό για να βρεθεί μια σύμβαστική λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα ακούμε τις ε, πολιτικές ομάδες. Σε αυτή τη φάση δεν δεχόμαστε μπλε κάρτα διότι δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η κυρία Κοσλόφσκα Ράγεβιτς. Δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Άκουσα όλα όσα υπόθηκαν και φαίνεται ότι όλοι συμφωνούμε. Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Κομισιόν όλοι υποστηρίζουν την οδηγία επιπλέον. Κανένα κράτος μέλος δεν αμφισβητεί τους στόχους της οδηγίας. Οπότε η ερώτησή μου είναι γιατί δεν έχει ακόμα τεθεί ενισχύ και γιατί σε κάποια κράτη-μέλη η παρουσία γυναικών σε εισηγμένες εταιρείε στα ΔΣ είναι μόλις 7%. Εάν ε, το επιχείρημα της επικουρικότητας ήταν σοβαρό, τότε τα κράτη-μέλη θα πρότειναν κάποιες λύσεις για να αλλάξει η κατάσταση. Γιατί δεν νομίζω ότι κανείς με κοινή λογική θεωρεί ότι η διαφορά 7 με 43% είναι κάτι το σωστό. Το ίδιο επίσης ε, και για τα υπόλοιπα ζητήματα είναι προφανές ότι δεν είναι ζήτημα ικανοτήτων. Άλλοι μηχανισμοί λειτουργούν. Πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτό κάποια αντίδραση πρέπει να υπάρξει. Εγώ στηρίζω αυτή την φανταστική οδηγία της Επιτρόπου, της κυρίας Ρέντινγκ, και έχει φτάσει πια η στιγμή οι ικανότητες να κρίνουν ποιος θα είναι διευθύνων ή διευθύνουσα σύμβουλος και ποιο θα είναι στο ΔΣ. Πρέπει να έχουμε σαφή κριτήρια και να αντιληφθούμε πώς ε, λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Δεν θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του ΔΣ να ορίζουν τους κολλητούς τους που τους ξέρουν χρόνια. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω της έλλειψης ε, υποδομών ε, για τα παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ισορροπία οικογενειακή και επαγγελματικής ε, ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να συγχαρούμε την Προεδρία για το αποτέλεσμα του διαλόγου που μόλις ολοκληρώθηκε και να στηρίξουμε την οδηγία στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ρέγνη, στους Δημοκράτες, δύο λεπτά. Μικρόφωνο, μικρόφωνο. Ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Χρειαζόμαστε ικανές, έξυπνες γυναίκες και άνδρες στην κεφαλή των ε, επιχειρήσεων, των ΔΣ. Πριν από 7 χρόνια, 7 χρόνια έφερε την πρόταση η Κομισιόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Διαπιστώσαμε ότι χρειαζόμαστε αντικειμενικά κριτήρια επιλογής και να είμαστε και πρακτικοί. Κοιτάμε τι γίνεται στις χώρες. Ποια χώρα έχει περάσει ανάλογους νόμους, ποια έχει κάνει πρόοδο με θελοντικά μέτρα. Δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδείχθηκε πάρα πολύ πρακτικό ότι χρειάζονται αντικειμενικά κριτήρια τα οποία μετά θα πρέπει να εφαρμοστούν. Δεν πάμε πουθενά με τον προαιρετικό χαρακτήρα. Χρειάζεται να είναι κάτι το υποχρεωτικό και με κυρώσεις. Η ισότητα είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει γίνει τόσο μεγάλη πρόοδος σε τόσες πολλές χώρες. Είναι δηλαδή κάτι το θαυμάσιο για τις επιχειρήσεις και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και τι συμβαίνει τώρα, πάρα πολλέ χώρες κρύβονται πίσω από τη νομική βάση. Ε, τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Είναι δεδομένη η νομική βάση, γιατί μόνο οι χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν επιτύχει καμία πρόοδο κρύβονται. Γι' αυτό ζητώ από την Ρουμανική Προεδρία την οποία χαιρετίζω καθώς επιτέλους ε, φέρνει αυτό το θέμα στο προσκήνιο να τραβήξει την κουρτίνα πίσω από την οποία κρύβονται κάποιες χώρες, χώρες όπως η Ουγγαρία που βλέπουμε τι γίνεται. Υπάρχει μάλιστα οπισθοχώρηση εκεί. Γι' αυτό ζητάω επιτέλους από την Προεδρία του Συμβουλίου να ζητήσει να μάθει αυτές οι χώρες επιτέλους τι έκαναν και να ψηφίσουν επιτέλους στο Συμβούλιο γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εδώ πέρα μια πολύ ισχυρή θέση, είναι ενωμένο και χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι επανήλθε επιτέλους αυτή η πρόταση. Βυσνιεύσκα, παρακαλώ για δύο λεπτά και να σέβεστε το χρόνο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύρια Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα Εάν δούμε τον δίκτυ ισότητας, βλέπουμε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα ΔΣ εταιριών. στις υψηλόβαθμες ε, θέσεις. Γιατί οι γυναίκες είναι ικανότατες, ε, έχουν προσόντα, θέλουν να δουλέψουν, είναι φιλόδοξες. σαφώς ε, δεν ε, έχουν λιγότερο ταλέντο γιατί λοιπόν τόσο λίγες γυναίκες ε, είναι σε αυτές τις υψηλόβαθμες θέσεις για εμένα ο βασικός λόγος είναι ότι η σταδιοδρομία τους εξελίσσεται με πιο αργό ρυθμό θέλουν όχι μόνο να τις εκτιμούν στη δουλειά αλλά και ως μητέρες Πρέπει να συνδυάσουν ε, την δουλειά με την οικογενειακή ζωή, θέλουν να γίνουν μητέρες, να φροντίζουν τα παιδιά τους. Γι' αυτό μένει πίσω η σταδιοδρομία τους. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα Δέλτα σίγμα. αλλά όχι με τεχνητό τρόπο, με οδηγίες. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να προτείνουμε λύσεις που θα δώσουν στις ε, γυναίκες την δυνατότητα να συνδυάσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Γιατί χρειαζόμαστε λύσεις ε, που θα μπορέσουν να εγγυηθούν αυτήν την ισορροπία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και θεωρώ ότι οι λύσεις αυτές προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι πολύ πιο επιτυχής. Η Eurostat μας λέει πως ε, το μισολογικό χάσμα διαφέρει πολύ ανάλογα με το κράτος μέλος, αλλά υπάρχουν χώρες όπου είναι πολύ ψηλό. Ευτυχώς η Πολωνία είναι μεταξύ των πέντε κρατών μελών ε, με το χαμηλότερο μισολογικό χάσμα και ευτυχώς ε, τελευταία έχουμε όλο και περισσότερες γυναίκες σε υψηλές θέσεις χωρίς να ληφθούν τέτοια τεχνητά μέτρα. Σας ευχαριστώ. Μπιλμπάο Μπαραντίκα, δύο λεπτά για την Άλντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλε τι προσπάθειε και για τη δέσμευσή σα για τι πρωτοβουλίε αυτέ. Βλέποντα το περιεχόμενο αυτών των ερωτήσεων και βλέποντα πώ έχουν φρακάρει στο Συμβούλιο αυτέ οι προτάσει για να υπάρξει ισότητα στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, θέλω να ζητήσω τρία πράγματα από τι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει. Συνέπεια, μακρόπνο όραμα και θάρρος. Πρώτα απ' όλα συνέπεια. Μα εδώ μας λένε συνέχεια για την ευφυή ανάπτυξη, για μια οικονομία που θα βασίζεται στο ταλέντο. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε το μισό ταλέντο που διαθέτουμε, που είμαστε εμείς οι γυναίκε, να μην φτάνει εκεί που μπορεί να βοηθήσει πιο πολύ. Στα διοικητικά συμβούλια, στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Ο, και όπω αποδεικνύουν όλες οι μελέτες αποδίδει περισσότερο. Εκεί θα επιτύχει, όπως το διαπιστώνουν όλες οι εμπειρίες που κάναμε σε ορισμένε όλες οι μελέτες που κάναμε σε ορισμένα κράτη-μέλη. Να έχετε το θάρρος να δείτε αυτή την πρόταση από την πλευρά της αποδοτικότητας. Εφόσον φοβάστε να το δείτε από την πλευρά της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ε, ίσης ευκαιρίας. Μακρόπνο όραμα τώρα. Η Ευρώπη είναι μία από τις περιοχές του κόσμου που προωθούν ε, πολιτικές ισότητας. Ας αξιοποιήσουμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Άλλες περιοχές ε, ασχολούνται τώρα με ιδέες που εδώ και χρόνια τις ε, προωθούμε. Ας κάνουμε το τελευταίο βήμα. Όπως είπαμε, όχι μόνο είναι δίκαιο και δημοκρατικό, αποδίδει, είναι κερδοφόρο. Όλα τα ωφέλη που θα ε, εξαγάγουμε από την πρόθεση αυτού του ταλέντου θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς. Επίσης, θάρρος. Πολλοί άνδρες σκέφτονται μόνο με αρσενικό τρόπο έναντι αυτού του φρακαρίσματος. να ξεπεράσετε τον φόβο σας, θα κερδίσετε. Είναι πολύ σημαντικό να ασχολείται κανεί με τα παιδιά, με του ηλικιωμένου. Είναι καταπληκτικό να έχει κανεί αυτή τη μαγική ευκαιρία να κάνει μια, έναν υπόθηκο δάνειο σε ένα σπίτι. Έτσι θα αξιοποιήσετε αυτό το τμήμα τη ζωή σα. Θα σα βοηθήσει να εξασκήσετε την συναισθηματική σα ε, νοημοσύνη. Θα σα συνδέσει με άτομα, με τι εμπειρίε, με τα προβλήματα, με τι ε, ευθύνε που αιώνε αποφεύγετε. Είμαι πεπισμένη ότι ένα κόσμο όπου και οι άνδρες θα αναλάβουν αυτές τις προκλήσεις θα είναι πολύ καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ. Ουρτασούν για τους πράσινους. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το διέξοδο για αυτή την οδηγία. Δεν έχει προωθηθεί το θέμα αυτό. Θα έπρεπε η Ρουμανική Προεδρία και το Συμβούλιο να προωθήσει αυτό το θέμα μέχρι το τέλος της θητείας. Γιατί όπως είπαμε έχει φρακάρει από το 2012. Θα πρέπει να υπάρχει 40% ποσόστοση για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο γιατί η οικονομική ισχύση είναι βασική για την ισότητα φίλων και έχει λειτουργήσει πολύ θετικά. Δεν τα επέλυσε όλα τα προβλήματα, αλλά στι επιχειρήσει που είναι στα χρηματιστήρια υπάρχει ψηλό ποσοστό γυναικών. Και δεν είναι θέμα όπου μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από την επικουρικότητα, όπω κάνουν πολλά κράτη-μέλη. Για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί η ισότητα φύλου είναι στόχο που αναφέρεται στι συνθήκε. Και η οικονομική δύναμη είναι βασικό θέμα για να υπάρχει ισότητα. Και δεύτερον, γιατί οι ανισότητες στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ορισμένε χώρε 7,4 μόνο, με 63% σε άλλε. Στα διοικητικά συμβούλια είναι τεράστια αυτή η ανισότητα, τεράστιο αυτό το χάσμα. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να επιτρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το χάσμα. Όπω είπαμε, η Νορβηγία είναι σίγουρα επιτυχία, δεν τα επέλυσε όλα και μπορούμε να, τα, να εξαγάγουμε ε, πορίσματα. Αλλά τα πορίσματα είναι τα εξή. Ένα είναι να είναι γυναίκε στα ειδικά συμβούλια, το βασικό όμω είναι να είναι και στι ανώτερε θέσει. Το να φτάσουμε στο πρώτο δεν σημαίνει πω επιτυγχάνουμε και το δεύτερο. Και αυτό που μα διδάσκει η εμπειρία τη Νορβηγία είναι ότι και η εφαρμογή δημιουργεί προβλήματα. Όμω από το 2013 το Κοινοβούλιο είπε να υπάρχουν κυρώσει για τι επιχειρήσει που δεν θα επιτυγχάνουν αυτού του στόχου. Για παράδειγμα, να μην συμμετέχουν στι δημόσιε προμήθειε, αν δεν έχουν φτάσει στο 40% που ανέφερε η οδηγία. Οπότε, είναι ένα βασικό τμήμα τη ε, νομοθεσία για να υπάρξει ισότητα. Εγώ θα ήθελα και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να επιχειρήσουν να μα στείλουν καλέ ειδήσει για το θέμα αυτό. Γιατί εμεί εδώ νομίζω ότι ομόφωνα σε αυτή την αίθουσα υποστηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Εκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί λοιπόν μόνο 24 ε, από τις 400 ε, θέσεις ε, στις ε, επιχειρήσεις στη Γερμανία που είναι στο χρηματιστήριο υπάρχουν γυναίκες και δεν υπάρχει καμία πρόεδρος. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε φτάσει σε κάτι καλύτερο. Αυτό είναι ντροπή. Και παγκόσμια δεν είναι καθόλου καλύτερη η κατάσταση. Από τις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις μόνο τρεις γυναίκες είναι επικεφαλής. Είμαστε στο 2019 και το συζητάμε ακόμη. Αυτό είναι ντροπή. Μας λέτε ότι είμαστε τόσο προοδευτικοί, αλλά υπάρχουν πολλοί που έχουν ε, ξεπερασμένες ε, αντιλήψεις ότι οι γυναίκες ε, πρέπει να είναι στο σπίτι ή σε χαμηλόμιστες δουλειές, ότι δεν είναι κατάλληλες λένε για τις ηγητικέ θέσεις στην οικονομία. Μα πόσο θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Αν δεν υπάρξουν δεσμευτικοί κανόνες, δεν θα επιτύχουμε τα ποσοστά που θέλουμε ε, για τι γυναίκε τα διοικητικά συμβούλια και τα υποπτικά συμβούλια. Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω συζητήσει. Ο κόσμο δεν είναι κόσμο των ανδρών. Είναι κόσμο για όλα τα φύλλα. Σε οποιοδήποτε φύλλο και να ανήκετε. Πρέπει να πούμε σε αυτού που είναι κατά των γυναικών και έχουν αναχρονιστικέ αντιλήψει ε, στι διοικητικέ θέσει ότι έχει περάσει η εποχή του. Παρακαλώ, Πάρκερ, για δύο μισή λεπτά. Η οδηγία για τι γυναίκε στο Διοικητικό Συμβουλίο όχι μόνο είναι προσβλητική, αλλά είναι και πατερναλιστική έναντι των γυναικών αυτών, οι οποίες κέρδισαν με το σπαθί τους και την αξία τους της θέση του. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία διαπιστώνει ότι έχει επιλεγεί μια ποσόστοση στη θέση τη και όχι μέσω λόγω των δεξιοτήτων της, αποδεικνύει ότι οι γυναίκες είναι κατώτερες και δεν μπορούν να επιτύχουν μόνο του την επιτυχία. Πώς ε, δικαιολογείται όμως η κατάσταση σε σχέση με τις γυναίκες που είναι σε χαμηλότερα επίπεδα των, ε, ε, της ιεραρχίας της επιχειρήσης και που δεν τις πρόχνει κανείς να πάνε πιο πάνω ή τα καταφέρουν μόνες τους. Είδαμε ότι και με την Ορβηγία ακόμα και στα συστήματα αυτά μόνο 7% των γυναικών έφτασαν στα διοικητικά συμβούλια. Αυτή η ιστορία με τις ποσοστώσεις πού θα σταματήσει. Πρώτα μιλήσατε για ποσοστώσεις για γυναίκες και άντρες. Μετά θα συνεχίσουμε πάντα με κατηγοριοποιήσεις και με ποσοστώσεις ατελείωτες. Για άλλη μια φορά, ακόμα περισσότερη παρέμβαση και επέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρώπη. Ναι, οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να βρουν μια δουλειά και να την κρατήσουν, αλλά εδώ επιβάλλεται μια σειρά από και απειλές και αυτό είναι μεγάλη απογοήτευση για τι επιχειρήσει. Ε, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα τι επιχειρήσει οι οποίε δεν καλύπτουν τι ποσοστώσει. Οι ποσοστώσει δεν λύνουν κανένα πρόβλημα ανισότητα. Και είναι πράγματι αντιπαραγωγικέ. Η γκρουπο 2.30. Πρόεδρε αυτή η φεμινιστική παράνοια βλέπω να συνεχίζεται. Τις γυναίκες θέλουμε να τις κάνουμε άντρε και τους άντρες γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω. Αρρώστια είναι, είναι τίποτα άλλο. Αλλά και ενώ κάποτε ήταν και φεδρό, όπως όταν ψηφίσαμε για το θέμα των γυναικών ε, στη γεωργία που δεν είναι αρκετές ε, οι βοσκοπούλες μπορεί να ήταν εφεδρό. Αλλά όταν μιλούμε για γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια των συγκεκριμένων επιχειρήσεων τότε γίνεται επικίνδυνο και ανοησία. Ας βγουν μερικοί άντρες να πούνε ότι είναι γυναίκες και έτσι καλύπτεται και το θέμα της ισορροπίας των φύλων. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό όμως και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Ε, βέβαια, όλη την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Κοινοβούλιο δίνει μόνο το τυποθήτο και τελικά είναι πολύ κακή η νομοθεσία. Και όσο πιο κακή είναι, τόσο πιο υπεύθυνο είναι και το Κοινοβούλιο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με νομοθεσία η οποία παρεμβαίνει στην οικονομική ελευθερία των επιχειρήσεων αλλά και στην εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Βλέπουμε διάφορες τέτοια, διάφορα τέτοια ψηφίσματα, ανόητα, παράλογα, άχρηστα να βγαίνουν από το Κοινοβούλιο. Πάντα όμως θα μιλάνε ή για μετανάστες ή για ομοφιλόφιλους ή για φεμινιστές που φαίνεται να είναι καλύτεροι από τους απλούς πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια αρρώστια. Ώρα να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν νομίζω ότι χωρεί μεταρρύθμιση και απευθύνομαι και στις άλλες χώρες. Ας ακολουθήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, ας βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας προετοιμαστούμε γι' αυτό και ας χτίσουμε μια νέα Ευρώπη όπως την είχαν οραματιστεί οι ιδρυτές που δεν θα παρεμβαίνει στην οικογενειακή πολιτική, δεν θα προσπαθεί να αλλάξει το ρόλο της γυναίκας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς θα πρέπει να κάνει τη διαχείριση μιας σωστής νομοθεσίας, μιας καλής νομοθεσίας σε περιορισμένο βαθμό. Και ελπίζω πραγματικά και εγώ να ζήσω να το δω αυτό, αυτή τη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω πει δυστυχώ εξ αρχή ότι δεν δέχομαι μπλε κάρτα. Σόσνιε, ένα λεπτό έχετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ να επιχειρήσω, κυρίε και κύριοι, να σα εξηγήσω κάτι. Σα παρακαλώ, α εστιάσουμε. Τα πορίσματά σα ε, είναι λανθασμένα, γιατί το σημείο εκκίνηση είναι λανθασμένο. Λέτε ότι οι γυναίκε έχουν ε, τα ίδια προσόντα, τι ίδιε ικανότητε με του άνδρε. Αυτό είναι εντελώ λάθο. Μετά διαμαρτύρεστε ότι δεν υπάρχει ίση εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια και σε θέσει λήψη αποφάσεων. Και θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία ότι υπάρχει κάποια πατριαρχική συνωμοσία που εμποδίζει τις γυναίκες από την ανάληψη τέτοιων ευθυνών. Αλλά κοιτάξτε, κοιτάξτε στην οικονομική δραστηριότητα. Αν οι γυναίκες δεν θέλουν να αναλάβουν τέτοιες ευθύνε. ή αν δεν θέλουν να απασχοληθούν καθόλου, είναι επειδή δεν έχουν ίσως τα προσόντα, ή επειδή δεν επιθυμούν μια τέτοια σταδιοδρομία. Ενώ, όπως ξέρετε, οι άνδρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες. Πώς θα τους ε, ε ανταμείψουμε για το γεγονό ότι πεθαίνουν ε, νεότεροι. Σας το λέει η αγορά. Οι γυναίκες δεν είναι σε αυτές τις θέσεις και δεν υπάρχει καμία συνωμοσία ανδρών. Ακούσαμε όλες τις πολιτικές ομάδες. Τώρα, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, οι ομιλητές, η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε. Ζούμε σε έναν κόσμο και σε μια κοινωνία όπου δεν είναι δυνατόν να αμφισβητείται η ισότητα ανδρών και γυναικών. Παρόλα αυτά, στα διοικητικά και εποπτικά συμβούλια δεν υπάρχουν επαρκεί γυναίκε. Οι γυναίκε είναι ο μισό πληθυσμό. Παρόλα αυτά, είναι πολύ λίγε σε αυτέ τι θέσει. Ε, ιδιαίτερα για τι επιχειρήσει ε, που είναι τι εισηγμένε. Στην Τσεχία, για παράδειγμα, είναι μόνο 9%. Ενώ οι γυναίκες σίγουρα έχουν τα ίδια προσόντα, τις ίδιες ικανότητες, αν όχι περισσότερες. Γιατί οι γυναίκες έχουν υψηλότερο ποσοστό, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και έχουν την ίδια φιλοδοξία. Παρά όλα αυτά δεν είναι επαρκής ο αριθμό των γυναικών σε αυτές τις θέσεις. Γιατί, Γιατί οι γυναίκες είναι πολύ σημαντικέ, ω μητέρε και για να φροντίζουν ε, τους ηλικιωμένους. Οπότε ξεκινάνε αργότερα τη σταδιοδρομία τους. Δεν θα βοηθήσουν οι ποσοστώσεις. Να προωθήσουμε και να επιταχύνουμε την σταδιοδρομία των γυναικών. Πρέπει να βοηθήσουμε τις ίδιες τις γυναίκες να μπορούν να συνδυάζουν την επαγγελματική με οικογενειακή ζωή. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Συμβούλιο επιτέλους να συμφωνήσει με αυτή την οδηγία ούτως ώστε επιτέλους να εφαρμοστεί ούτως ώστε αυτή η οδηγία να βοηθήσει τον συνδυασμό της ε, επαγγελματική και οικογενειακής ζωής. Επιτέλους να γίνει, να εγκριθεί και να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Και σας ρωτώ, τι εμποδίζει τα κράτη-μέλη μέσω της δικής τους ε, νομοθεσίας να προωθήσουν την ισότητα των γυναικών. Για παράδειγμα, η Ισπανία. Πιστεύω ότι αυτό που έκανε η Ισπανική κυβέρνηση μπορεί να το κάνει και σε εθνικό επίπεδο. Να αποφασίσει εγώ ω χώρα θα προωθήσω αυτά τα μέτρα που επιχειρώ να προωθήσω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όποιο θέλει μπορεί να το κάνει. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Και φυσικά και η Ένωση μπορεί να δώσει καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ, Γκούτερλεντ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πάνω από το 65% των πτυχιούχων είναι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν τις γνώσεις για να καταλάβουν τις ε, κορυφαίες θέσεις στα ΔΣ. Και όμως ακόμα ε, δεν το κάνουν. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι μόνο άδικο, είναι και βλακώδες. Σημαίνει ότι χάνουμε γνώση. Δεν υπάρχει καινοτομία. Ε, βλέπουμε ότι σε πολλές εταιρείες οι γυναίκες είναι πολύ πιο καινοτόμες από τους άνδρες και οι εταιρείε που έχουν περισσότερες ε, γυναίκες από άνδρες ε, παρέχουν ε, πολύ καλύτερες δυνατότητες για τις εταιρείε αυτές. Παρόλα αυτά, πολλές εταιρείε και πολιτικοί εξακολουθούν να μάχονται αυτήν την ιδέα ότι τουλάχιστον 40% των μη εκτελεστικών μελών θα πρέπει να είναι από το φύλλο που εκπροσωπείται. Γι' αυτό ακριβώς είναι περίεργο να βλέπουμε την Ισπανία να μεταβάλει στάση στο Συμβούλιο. Δεν θέλουμε άλλα ωραία λόγια. Θέλουμε επιτέλους να γίνει κάτι στην πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τις ε, γυναίκες στα Δέλτα Σίγμα, ας δούμε εδώ πέρα τι γίνεται σε Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν. Είχαμε 12 πρόεδρους ε, της Κομισιόν, καμία γυναίκα. 30 πρόεδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μία γυναίκα και 78 πρόεδρους του Συμβουλίου, σε νέα γυναίκες. Λοιπόν, ε, γιατί δεν ε, το βλέπουμε, γιατί δεν ζητάνε συγγνώμη οι άντρε ε, πρόεδροι για αυτό το γεγονός. Δηλαδή χρειάζεται πραγματικά οδηγία. Όλοι είναι ίσοι ε, ενώπιον του νόμου, στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία. Έτσι τα έχουμε ρυθμίσει στο Σύνταγμα της Πολωνίας. Έχουμε μια κοινωνία στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση, γιατί είμαστε όλοι ίσοι. Ε, ενώπιον του νόμου. Αυτή είναι η εντολή και πρέπει να την σεβόμαστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπέτσερα Μπαστερετσέα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας κύριε Επίτροπε και για την αποφασιστικότητά σας. Σήμερα ορισμένοι λένε ναι. ότι οι γυναίκες δεν είναι σε τέτοιες ηγετικές θέσεις γιατί δεν το επιδιώκουν. Όμως το ποσοστό γυναικών ε, των εισηγμένων ε, ευρωπαϊκών εταιρεών από 10% το 2005 πέρασε στο 22% το 2015. Άρα κάτι γίνεται. Ορισμένοι λένε ότι δεν χρειάζεται, εφόσον αλλάζει η κατάσταση η πρωτοβουλία αυτή για την ίση εκπροσώπηση. Όμω οι γυναίκε ε, είναι επικεφαλεί μόνο στο 7% των εισηγμένων και μόνο το 6% ε, στις κυριότερες επιχειρήσεις. Ε, εξακολουθεί να υπάρχει η γυάλινη οροφή. Υπάρχουν εμπόδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση. Για να γίνει αυτό πρέπει το Συμβούλιο να προωθήσει αυτήν την οδηγία. Η ίση εκπροσώπηση είναι θετική για όλους, για τις επιχειρήσεις, για τις γυναίκες. Οι επιχειρήσεις που έχουν γυναίκες έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να ε, καταλάβουμε ότι είναι το πιο λογικό να υπάρχει αυτή η ισότητα. Πρέπει να προχωρήσει αυτή η οδηγία, να αναλάβει την ε, προώθηση αυτής της ιδέας που απαιτούν οι Ευρωπαίοι και ελπίζω η Ρουμανία να παίξει το ρόλο της. Κυρία Φορέντσα, για ένα λεπτό, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, των ε, Πρασίνων και των Σοσιαλιστών Δημοκρατών που κατέθεσαν αυτή την προφορική ερώτηση, τις προφορικές ερωτήσεις σε σχέση με την ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων ε, και με την συνσηγήτρια έχουμε εργαστεί προς την κατεύθυνση. Θα ήθελα να επισημάνω ωστόσο ότι εδώ αντιμετωπίζουμε, κοιτάμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύμπτωμα αυτής της διακριτικής μεταχείρισης. Εδώ θα έπρεπε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τις εξελίξεις αυτές που μπορεί να οδηγήσουν σε περισσότερες ακόμη διακρίσεις. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει λοιπόν απαντήσεις αποφασιστικές όχι μόνο για αυτή την ε, γυάλινη οροφή που αφορά τις γυναίκες και επιτρέπει μόνο στο 1% να την ξεπεράσουν, σε όλες τις ε, διακρίσεις βάρος τους και εις βάρος ουδήποτε, είτε πρόκειται για φίλο, φιλή, ε, προέλευση λοιπά Πρέπει να καταπολεμείται κάθε διάκριση και πρέπει το Κοινοβούλιο να δώσει ένα έναυσμα σοβαρό προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους λοιπόν που καταθέσαν τις προφορικές ερωτήσεις, αλλά βλέπω ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και όπως υπενθύμησε και η κυρία Ορτασούν, θα μπορούσε, θα, είχε, θα μπορούσε η περίοδος η βουλευτική αυτή να είχε κάνει πολύ περισσότερα ε, για τα θέματα της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η κυρία Γιούτο για ένα λεπτό. Ε, το 2012, χρόνια πριν, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια πρώτη πρόταση για σχέδιο οδηγίας ε, για τις θέσεις των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων που έμεινε σε αδιέξοδο στο Συμβούλιο για στόχο είχε να εξασφαλίσει περισσότερη ισότητα στις, ε, στην παρουσία των γυναικών, ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Βέβαια ξέρουμε ότι αυτό αυτή η ισότητα, ο στόχος της ισότητας μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο όταν στο πεδίο της δράσης μπορούμε να αποδείξουμε την αξία μας, την αξία μας, τις δεξιότητες μας που εμείς οι γυναίκες έχουμε και θέλω να διαβεβαιώσω τον συνάδελφο, λυπούμε βέβαια για λογαριασμό του, αλλά είναι αποδεδειγμένο πως οι γυναίκες έχουν και περισσότερα πτυχία και δεξιότητες προς από τους άντρες ε, και τα, το σημείο εκείνης αυτής της οδηγίας και των προτάσεων που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ενισχυτικές διαπιστώσεις γιατί μόνο 13,20% κατελάμβαναν στις υψηλές θέσεις γυναίκες και εδώ θέλω να ρωτήσω τη Ρωμανική Προεδρία τι είδους μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να ε, σπάσει αυτή τη γυάλινη οροφή επιτέλους και εάν σκοπεύει να καταστεί εκπρόσωπος της φωνής των γυναικών, εσείς κυρία Υφυπουργέ, εκπρόσωπος της φωνής των γυναικών στο Συμβούλιο. Ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γνωστό ότι οι άντρες υπερεκπροσωπούνται στα ΔΣ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα, το 2017 οι γυναίκες ήταν μόλις το 1 τέταρτο των μελών των ΔΣ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιριών στην Ένωση. Το 2015 υπήρχαν περισσότεροι ε, Δέλτα Σίγμα, ε, περισσότεροι, με συγχωρείτε, διευθύνοντες ε, σύμβουλοι που λεγόταν Τζον παρά γυναίκες. Λοιπόν, ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο το ΔΣ. Από εκεί θα διαχυθεί σε ολόκληρη την ε, ιεραρχία. Ε, οι γυναίκες συχνά βρίσκονται σε άλλους ρόλους εντός των εταιριών, ενώ οι άντρες βρίσκονται σε θέσεις οι οποίες θεωρούνται πιο σοβαρές. Οι γυναίκες είναι στο ανθρώπινο δυναμικό, δημόσιες σχέση κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να αντικατοπτρίζονται ολόκληρε όλες οι απόψεις ε, που υπάρχουν στην ε, κοινωνία. Αλλιώς ε, συνεχώς αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα ΔΣ θα προάγουν τους ομοίους τους. Δηλαδή αν υπάρχουν ήδη περισσότεροι άντρες θα προάγονται περισσότεροι άντρες. Αυτό δεν έχει νόημα. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μια τέτοια πρακτική θα προωθούσε αυξημένη παραγωγικότητα και ισότητα στα εισοδήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κοφεράτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συχνά στις συζητήσεις μας ε, επενθυμίζουμε ότι η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά βέβαια στη συμπεριφορά, την πρακτική, έχουμε διαφορετικό προσανατολισμό, όπως άλλωστε αποδεικνύει και η σημερινή συζήτηση. Αυτό που κάνει το Συμβούλιο είναι πονίδιστο πραγματικά, γιατί βρισκόμαστε ενώπιον μιας οδηγίας που έχει με ευρύτατη πλειοψηφία εγκριθεί πριν 10 χρόνια και περισσότερο και δεν έχει προχωρήσει ούτε βήμα το Συμβούλιο. δεν πρόκειται για κάτι το εξαιρετικά απαιτητικό ή ρηξικέλευθο αυτό που στάει η οδηγία. Ένα 40% για παρουσία των γυναικών, μια αντίστοιχη ποσόστοση για τις ε, θέσεις ε, της ε, ιεραρχίας παραμένει ανοιχτό το θέμα εξάλλου και της ισότιμης ε, αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και αυτό που ζητούσαμε εμείς ήταν ένα μικρό βήμα, ένα μικρό βήμα προς σωστή κατεύθυνση που θα επέδεικνει μόνο απλώς καλές προθέσεις. Ελπίζω το Συμβούλιο να επιδείξει τη βούληση και να αποδείξει ότι σκοπεύει να το κάνει, να αλλάξει προς την ορθή κατεύθυνση, δηλαδή να δείξει σεβασμό και να ε, προωθήσει και την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κούνεβα, ένα λεπτό σε μια κοινωνία χωρίς ισότητα αλήθεια τι αρμονία και τι ομορφιά μπορεί να επικρατήσει αναρωτιόταν ο Τζον Μίλτον. Το ίδιο αναρωτιέμαι και εγώ. Το γυάλινο ταβάνι που εμποδίζει την σταδιοδρομία χιλιάδων εργαζομένων γυναικών ανατρέπει τις ζωές τους. Εργαζόμενες με εμπειρία, σποντές και κατάρτιση αποκλέονται από διευθυντικές θέσεις αμείβονται λιγότερο τιμωρούνται αν έχουν ή αν θέλουν οικογένεια δέχονται παρενοχλήσεις διάφορων μορφών. η πρόταση οδηγίας είναι σίγουρη, σίγουρα μια ακόμα ευκαιρία να διορθώσουμε ανισότητες που επικρατούν. όμως γιατί αργεί η υιοθέτησή της; ρωτώ το συμβούλιο ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο του τα ταβανιού στις επιχειρήσεις και πώς σκοπεύει να προάγει την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της ρωμανικής προεδρίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κούνεβα. Ο κύριος Ντουαχμαχτάν δεν είναι εδώ και έτσι προχωρώ στη διαδικασία Catch Παρακαλώ με προσοχή στο χρόνο. Κίνηση, ένα λεπτό. Έλα Κατερίνα. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Το 2017 ήταν ένα τέταρτο μόνο των μελών των, συμβουλίων, των διοικητικών συμβουλίων των εισηγμένων στα χρηματιστήρια ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι γυναίκες και όμως ακόμα τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ε, στα, στην εκπροσώπηση του στα διάφορα κράτη μέσα στην Ένωση. Οι ικανότητες βεβαίως των γυναικών είναι αμφισβήτητες και οι δεξιότητες τους. Είναι παράδεκτη λοιπόν αυτή η διάκριση εις βάρος τους για λόγους στερεοτύπων που ταυτόχρονα όμως ε, προξενεί προβλήματα και στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσει μια καλύτερη ισότητα φύλων, εκπροσώπηση των φύλων η πιο ισόρροπη, χρειάζεται να εισαχθούν και νομοθετικά μέτρα. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Έστω και με ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών. Έγινε στην πατρίδα μου την Ιταλία παραδείγμα κάτι μια τέτοια πρωτοβουλία η οποία έφτασε να, να εξασφαλίσει πάνω από το 33% των ε, γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και έτσι να, υπάρχουν πολύ καλύτερη, να υπάρχει πολύ καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών. Καλό λοιπόν τη Ρουμανική Προεδρία το ταχύτερο δυνατό να εξασφαλίσει πρόοδο για την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων επιχειρήσεων. Η κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό το συζητάμε εδώ και 7 χρόνια. Το είπαν όλοι οι συνάδελφοι. Εγώ θέλω να απευθώ κυρίω στου άνδρες που αναφέρθηκαν σε ανισότητες. Γιατί υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι δουλεύουν στο σπίτι και αισθάνονται μειονεκτικοί. Ε, κοιτάξτε, οι γυναίκε ε, και βιολογικά είναι παντού οι καλύτερε. και στις ε, επιχειρήσει και στο σπίτι γιατί περισσότερε έχουν ούτω ή άλλω δύο δουλειέ και μια επαγγελματική δραστηριότητα και κάνουν τη δουλειά στο σπίτι και είναι καλύτερε για τα δικαιωτικά συμβούλια μπορούν να κάνουν δύο πράγματα την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν επαγγέλματα που είναι μόνο για άνδρες ή μόνο για γυναικέ και ελπίζω κυρία Υπουργέ και κυρία Επίτροπε να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή την ε, ε, μειοψηφία άρνηση κυρία στο Συμβούλιο. Λυπάμαι που πρέπει να υπάρχουν ε, ποσοστό, αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Αν η κοινωνία δεν καταλαβαίνει πώ πρέπει να προωθηθούν οι γυναίκε, πρέπει να παρέμβουμε. Συμφωνώ, κύριε Επίτροπε, η οδηγία για, την, ε, ε, για το συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματική ζωής και όλα τα άλλα που είπατε, όλες οι μελέτες το αποδεικνύουν, όλα αυτά πρέπει να γίνουν πραγματικότητα γιατί θα κερδίσει η κοινωνία. Ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Γυναικών και στην κοινωνία και στις ε, βασικές θέσεις και στην οικονομία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και προφανώς πρέπει αυτό να αλλάξει. Και φυσικά θα πρέπει οι γυναίκες να εκπροσωπηθούν και στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Αλλά η κοινωνική μηχανική, το social engineering το οποίο επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι μπορεί να πετύχει στον τομέα αυτό. Ούτε μπορεί να αναγκαστούν οι επιχειρήσεις να κάνουν κάτι διαφορετικό. μπορεί όμως η ευρωπαϊκή ένωση να κάνει κάτι άλλο και επειδή είναι εδώ και ο κύριος juncker και ακούω λέω το εξής 140 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ο προϋπολογισμός της ευρωπαϊκής ένωσης 70 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων 2,5 τρισεκατομμύρια έχει δώσει ο κύριο ντάγκη λέω λοιπόν να μην γίνεται καμία χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια ούτε από δάνεια ούτε να αγοράζονται ομόλογα από την κεντρική τράπεζα εάν οι συγκεκριμένε επιχειρήσει δεν έχουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. να δείτε πώ αμέσω μόνε του οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν και θα αλλάξουν την τακτική και θα έχουν την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια διότι δεν θα έχουν πρόσβαση ούτε στην οικονομία ούτε στα ομόλογα ούτε βεβαίω στα χρήματα που είναι και από το ε, πρόγραμμα juncker. με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια απάντηση και αναγκάζουμε τις επιχειρήσεις να έρθουν σε αυτά τα οποία εμείς επιθυμούμε. ευχαριστώ. Σας παρακαλώ να είμαστε όλοι αυστηροί με το χρόνο. Από εδώ και μπρος όποιος ξεπερνάει το λεπτό του θα ε, χάνει το μικρόφωνο. Σπίνα παρακαλώ. Πρόεδρε, ναι, αυτή η συζήτηση σήμερα νομίζω δείχνει μια μεγάλη σύγκληση του Κοινοβουλίου προς την υποστήριξη της ε, οδηγίας αυτής και σας παρακαλώ προσέξτε το δεν λέει τίποτε το καταπληκτικό ένα μικρό βήμα που όμως πάει προς σωστή κατεύθυνση γιατί δεν επιβάλλει την παρουσία των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εδώ αυτή η οδηγία. Απλώς καταγράφεται πως δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπείται μόνο το 50% δηλαδή ο ανδρικός κόσμος στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων των εισηγμένων και ότι χρειάζεται και η εκπροσώπηση των γυναικών. Μια πραγματικότητα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι όπως πάντα το Συμβούλιο και το λέω αυτό με μεγάλη πικρία αλλά και μεγάλη ανησυχία διότι βλέπουμε εκεί μία στάση. Έχουμε από τη μία πλευρά μια στάση του Κοινοβουλίου που θέλει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποια βήματα προόδου. Ενώ από την άλλη έχουμε τη συμπεριφορά και στάση του Συμβουλίου και, που το οποίο δυστυχώς πολύ συχνά, Πρόεδρε, παρεμποδίζει αποφάσεις και επιλογές που βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως και η προτεραιότητα πρέπει να είναι αυτή η ισότητα και χρειάζεται δράση. Ευχαριστώ πολύ. Σμαέσνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για αυτήν την οδηγία και για την συζήτηση για διάφορους λόγους. Είναι καλό το ότι συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άντρες γιατί πρέπει από κοινού να επιτύχουμε την ισότητα για τις γυναίκες και την εκπροσώπησή τους σε όλους τους ε, τομείς γιατί είναι αρκετά καλές ε, όσο και οι άντρες και αναφέρθηκε το μισθολογικό χάσμα ξέρω ότι στη Γερμανία είναι υψηλότερο από σε άλλες ε, χώρες συζητάμε ήδη σε μας ένα νόμο περί ισότητας με διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποια κράτη-μέλη έχουν τέτοιους ε, νόμους για το φύλλο που υποεκπροσωπείται. Είναι κρίμα το ότι το συζητάμε ακόμα. Έπρεπε να υπάρχει ήδη. Και χαίρομαι που η συναρφός Ρέγνερ λέει ότι είναι επιτέλους το ευρωπαϊκό DNA. Γι' αυτό ελπίζω να υπάρχει ευρεία στήριξη και να καταλήξουμε κάποτε σε ένα αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ η κυρία Ward για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Είναι εκπληκτικό να βλέπουμε πως η πρωτοβουλία αυτή για την ισότητα μπλοκάρει στο Συμβούλιο μετά από πέντε χρόνια. Πραγματικά δείχνει πόσο συντηρητικές είναι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Είναι ανησυχητικό το ότι είναι τόσο αμφιλεγόμενη αυτή η πρωτοβουλία. Και βλέπουμε ότι βεβαίως η ισότητα, αν και είναι σημαντική κυρίως, απευθύνεται σε προνομιούχες γυναίκες και δεν ασχολούμαστε με τις μη προνομιούχες. Στον κόσμο των επιχειρήσεων οι γυναίκες υφίστανται πολλές διακρίσεις. Αντιμετωπίζουν φοβερές προκλήσεις. Μαύρες, Ρωμά, μετανάστες, ανάπηρες, ε, ξεχνιούνται και στην πολιτική και στις επιχειρήσεις μετά από την συμφωνία που επετέφθη την προηγούμενη εβδομάδα στην οδηγία για την ισορροπία οικογενειακής ε, και επαγγελματικής ζωής ζητάω από την Προεδρία να επιτύχει επιτέλους μια συνένεση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Μιράντα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση εδώ που επικρατεί στο Συμβούλιο νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική. Αρκεί να δούμε μια φωτογραφία του Συμβουλίου. Λίγες οι γυναίκες στο διοικητικό, στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Στην ε, Σουηδία το πολύ να φτάσουν στο 36%. Όμως είναι πολύ μακριά τα ποσοστά αυτά από τα επίπεδα που ζητεί η οδηγία. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, σε προηγούμενη σύνθεση του Κοινοβουλίου, το ίδιο θέμα. Και δυστυχώ βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση πάντα και δεν γίνονται σεβαστέ οι οδηγίε. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία παρέμβαση. Dear President, dear Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, εγώ ως ε, ε, Ευρωβουλευτή από την Ρουμανία, καλωσορίζω το γεγονό ότι αυτή η οδηγία είναι μία από τι προτεραιότητε τη Προεδρία μου για την ισότητα των φύλων. Σε κάποια κράτη-μέλη άλλαξε η κατάσταση πρόσφατα και ε, έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση για το θέμα αυτό. Ο λόγο υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικέ θέσει ε, είναι περιπλοκο Υπάρχει βεβαιω η νοοτροπία που υπάρχει και σε διοικητικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Η Γιάννη οροφή στην οτροπία των επιχειρήσεων όχι μόνο υποτιμά την συμβολή των γυναικών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, αλλά αποθαρρύνει και τι γυναίκε από την προσπάθεια να προωθήσουν τη σταδιοδρομία του και να αναπτύξουν τι δυνατότητέ του στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η δική μου εμπειρία μου επιτρέπει να σα πω ότι οι γυναίκε όταν αναλαμβάνουν την ηγεσία κάποιων επιχειρήσεων προσθέτουν αξία και αυξάνεται η επιχείρηση, κάνει καλύτερε προτεραιότητε για, για τι ανάγκε των γυναικών και αλλάζει την οτροπία τη επιχείρηση. Εκφράζω λοιπόν τη στήριξή μου για τι προσπάθειε Ρουμανική Προεδρία ούτως ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση για αυτή την οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, έκλεισε η συζήτηση. Για να απαντήσει τώρα η κυρία Γιούροβα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ για την αποφασιστικότητα και την στήριξη του Ευρωπαϊκού του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, όπως φάνηκε στην συζήτηση και χαιρόμαι που υπάρχει και ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Θα ήθελα να καταλήξω λέγοντας ε, λίγα λόγια. Πέρα από την σαφή στήριξη της Κομισιόν που ήδη εξέφρασα, θα ήθελα να σας πω πως ε, δεν ε, περιμένουμε να ξεμπλοκαριστεί το θέμα αυτό στο Συμβουλίο, γιατί υπάρχει πολλή δουλειά που μπορεί να γίνει για να στηρίξουμε την ε, μεγαλύτερη ισότητα ε, όχι μόνο στον κόσμο των επιχειρήσεων. Θα ήθελα και πάλι να αναφέρω κάποια στατιστικά στοιχεία. Οι γυναίκες είναι πάνω από το 50%. 62% των πτυχιούχων. Οπότε θα έλεγε κανείς πως ε, το φυσιολογικό θα ήταν να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση των γυναικών σε διάφορους τομείς. Ας συγκρίνουμε τους αριθμούς όμως. Έχουμε 22% γυναικών στα ΔΣ. Μόλις 6% των ε, διευθυνόντων των συμβούλων. 20% γυναικών βουλευτών. Έχουμε κάποιες ε, κυβερνήσεις ε, στα κράτη-μέλη με μία ή δύο γυναίκες. Προσφάτως είχαμε κυβέρνηση χωρίς γυναίκα. Ας δούμε τώρα τα θετικά παραδείγματα. Στην ε, Κομισιόν ήδη φτάνουμε το 40% στις θέσεις τις διευθυντικές. Μια πολύ έξυπνη διαδικασία η οποία εγγυάται τον ε, δίκαιο ανταγωνισμό χωρίς ε, προκαταλήψεις ε, που βλέπουμε αλλού και χωρίς εμπόδια. Και να αντιδράσω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Ζόλταξ. Ε, με, ε, ως γυναίκα εντός κομψιών, δεν χρειάστηκε να γίνω άντρα για να φτάσω σε αυτήν την θέση και να συνεισφέρω στην λήψη των αποφάσεων. νομίζω πως κατά σύμπτωση είναι εδώ και ο Ζαν Κλοντ αλλά ε, υπάρχουν τουλάχιστον 9 γυναίκες στην Κομισιόν και όλοι οι συνάδελφοι νομίζω κάνουν ε, πολύ σωστή δουλειά με το να μεταφέρουν την οπτική των ε, γυναικών στην λήψη των αποφάσεων. Όταν συγκρίνουμε αυτούς τους αριθμούς λοιπόν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Γι' αυτό ακριβώς ε, εργαζόμαστε σκληρά για να το αλλάξουμε. Και δεν ε, περιμένουμε μόνο... Δεν ξεμπλοκάρουμε μόνο αυτή την οδηγία. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κυρία Πάρκερ, να διαβάσετε την ε, τωρινή εκδοχή της οδηγίας. Τίποτα δεν λέει ότι το μόνο προσόν είναι να είναι κανείς γυναίκα. Ζητάμε απλά δίκαιο ανταγωνισμό και συνεργασία. Καλό είναι να ε, δείτε την ε, τελευταία έκδοση την οποία προωθούμε. Αυτή τη στιγμή ήδη τα μισά κρατημέλη έχουν σχετική νομοθεσία, οπότε πρόσεχος θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Και γεγονός είναι ότι τα κρατημέλη μπορούν να δράσουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να περιμένουν να ξεμπλοκάρει η οδηγία γιατί από αυτά εξαρτάται να κινηθούν. Εν τω μεταξύ η Κομισιόν δεν περιμένει κάνουμε και μη νομοθετικό έργο, στηρίζουμε την ε, χάρτα της ποικιλομορφίας, ε, την οποία έχουν συνυπογράψει 10.000 ε, μεταξύ των οποίων μεγάλες εταιρείες, η IBM, Siemens, πολυεθνικές, που προωθούν την ιδέα αυτή η οποία είναι υποφελής ε, για τις επιχειρήσεις ε, πολλά κρατημέλη ε, και όπου δεν υπάρχει νομοθεσία εξάγουν και διαδίδουν αυτό το θετικό μήνυμα. Χρηματοδοτούμε και πολλά έργα τα οποία προωθούν ακριβώς την ποικιλομορφία. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο Β αν θέλετε να μην ε, περιμένουμε την νομοθεσία κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα αλλά θα ήθελα να επαναλάβω πώς ε, θεωρούμε πως ε, θα εγκριθεί τελικά αυτό το νομοθέτημα και πάλι θα ήθελα να επαναλάβω ότι ελπίζουμε ότι η Ρουμανική Προεδρία θα κάνει πολύ καλή δουλειά σας ευχαριστώ η κυρία Τσότ για το Συμβουλίο Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε, και κύριοι. ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Όπως είπα και στις αγωγικές μου παρατηρήσεις, η προσήλωση του Συμβουλίου στην ισότητα των φύλων είναι πραγματική και απαρασάλευτη. Η Προεδρία της Ρουμανίας οργανώνει διμερείς συνομιλίες με την ανασχετική μειοψηφία για να αναζητήσει δυνατότητες λύσης. Έχουμε σχεδιάσει ακόμη ε, συνεδριάσεις σε επίπεδο ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό. Δεν πρέπει όμως και να λησμονούμε ότι η Προεδρία είναι στα χέρια και υπό τον έλεγχο των κρατών μελών. Απαιτείται λοιπόν μια ειδική πλειοψηφία για την ε, πρόθεση αυτού του έργου. Ε, επιπλέον των όσων έχουμε κάνει σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να προαγάγουμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πάντως, όπως είπα και νωρίτερα, προετοιμάζουμε και μια σειρά συμπερασμάτων για την ε, διαφορά στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις πολιτικές ε, συγκερασμού του οικογενειακού και του επαγγελματικού βίου. Ελπίζουμε ότι αυτά τα συμπεράσματα θα ε, εγκριθούν στο Συμβούλιο Αψικός στις 13 Ιουνίου και θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι η Ρουμανική Προεδρία θα υποδεχθεί στο Βουκουρέστι το Φεβρουάριο την ε, ομάδα εργασία για την ε, ισότιμη εκπροσώπηση, για την ενσωματωστία σα του φίλου καλύτερα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δούμε και τους υπουργούς ε, τους αρμόδιους Αψκό στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα σήμερα εδώ με την κοινή δουλειά του, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να θέσουν ένα τέρμα στην, στις διακρίσεις και την αδικία και να εξασφαλίσουν ε, ως πραγματικότητα για όλες τις γυναίκες και τους άντρες την ισότιμη μεταχείριση σε μια περίοδο μετάβαση, σε μια περίοδο κλειδονισμών όπου αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Το μέλλον όμως είναι η ισότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ την κυρία Σότ και τώρα ολοκληρώνεται έτσι η κοινή συζήτηση. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Φινλανδίας για το μέλλον της Ευρώπης. Κάνουμε μια διακοπή ενός λεπτού. Καταρχάς θέλω να ευχαριστώ τον Φιλανδό, τον Φιλανδό Πρωθυπουργό που είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε τις διαφορετικές θέσεις των, διαφορετικών, των διάφορων χωρών ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επισημάνει δύο-τρία περισσότερα σημαντικά θέματα και θέλουμε περισσότερε εξουσίε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Θέλουμε να ενισχύσουμε και όχι να καταστρέψουμε την Ευρώπη. Στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θέλουμε την αλλαγή από το 1,1 στο 1,3 του όγκου του. Έχουμε επίσης ε, προτίμηση για τους ιδίους πόρους. Ε, μετανάστευση είναι πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμιση των κανόνων του Δουβλίνου και θέλουμε να δούμε απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εχθές και σήμερα στο επίκεντρο των συνομιλιών μας μάλιστα έθεσαμε δύο κέρια ζητήματα, το Brexit και τη Βενεζουέλα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για μα να ενημερωθούμε για τις ιδέες σας. για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ξέρουμε ποιες είναι οι θέσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ποιε είναι οι θέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίως, τα κράτη-μέλη έχουν το καθένα τι δικέ του θέσει και τώρα είναι σημαντικό να ακούσουμε ποιε είναι οι θέσει τη Φιλανδία. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να δώσετε τώρα τις, ε, το, να εκδηλώσετε τον ενδιαφέρον σας για το Catch the αμέσως μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Θα κλείσουμε τον κατάλογο των αγορητών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας φέρνω τους χαιρετισμού από την πολύ κρύα Φιλανδία. Είμαι στη Βόρεια Φιλανδία την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί μένω, η θερμοκρασία ήταν μείον 30 και είχαμε ένα μέτρο περίπου χιόνι. Έχουμε βαρύ χειμώνα. Ε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στα πλαίσια των ε, πολύ δύσκολων καταστάσεων. Οι συζητήσει για το μέλλον τη Ένωση είναι ουσιώδει για δύο λόγου. Πρώτα απ' όλα, για να εκπληρώσουμε το όραμα τη διακήρυξη τη Ρώμη, πρέπει να συζητήσουμε πώ θα επιτύχουμε επαρκή ενότητα για να λαμβάνονται αποφάσει και να εφαρμόζονται. Δεύτερον, πρέπει να συζητήσουμε για να διαπιστώσουμε τις ε, προτεραιότητες των ΜΕΝ και των ΔΕ για τη δράση και τον προπολογισμό της Ένωσης. Οι χώρες της Ένωσης είναι κάτι που γνώρισα όταν ήμουν επιχειρηματίας. Είχαμε θηγατρικές σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Όταν ήμουν 30 και κάτι, θυμάμαι ότι ταξίδευα για να συναντήσω τον επικεφαλής μιας μεγάλης ε, γαλλικής εταιρείας. Στο αεροπλάνο διάβασα έναν ταξιδιωτικό οδηγό που, είχε, που είχε δανειστεί η γυναίκα μου από, ένα, από μια βιβλιοθήκη. Έλεγε ότι δεν θα πρέπει ποτέ να κάνεις ερωτήσεις για την οικογένεια όταν ε, ε, συναντάς ένα Γάλλο για επαγγελματικού λόγους. Όταν έφτασα στην ε, συνεδρίαση, στην, συγγνώμη, στο δείπνο, ο επικεφαλής ήταν με τη γυναίκα και την κόρη του και η πρώτη ερώτηση που μου έκανε ήταν πες μου για την οικογένειά σου. Τότε κατάλαβα ότι εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε πολλά κοινά και μπορούμε να συνοηθούμε. Έχουμε περισσότερα κοινά από όσα νομίζουμε. Ήδη το 1920 ο ιδεολογικός πρόδρομος και ιδρυτής ε, του κεντρικού κόμματος του κέντρου της, Φινλανδία, Φινλανδίας, ο Σάντρι Άλκιο, έγραψε ότι για να υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη, η Ήπειρος θα πρέπει να οδηγηθεί προς τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης. Ανέφερε ακόμη και ένα κοινωνόμισμα. Ήταν πρωτεργάτης από πολλές ε, απόψεις. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, η διεθνή συνεργασία και η προώθηση της ειρήνης και της οικονομικής ανάπτυξης έχει υπάρξει φάρος για τη Φιλανδία. Αγαπητοί φίλοι, τα τελευταία χρόνια όμως ε, είδαμε πολύ λαϊκισμό στην Ευρώπη. Είδαμε τι συμβαίνει όταν, και που οδηγεί ο λαϊκισμός, όταν προτείνονται υπεραπλουστευμένες λύσεις για περίπλοκα θέματα. Στο τέλος κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό συνέβη και στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα αποτελέσματα είναι ενώπιον όλων μας. Αλλά δεν είναι μόνο το Brexit, όπου βλέπουμε τα αποτελέσματα του λαϊκισμού. Βλέπουμε ότι μειώνεται το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτά δεν θα τα περιμέναμε. Στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει τις κοινέ αξίες της μέσω της εξωτερικής της πολιτικής αν δεν μπορεί να τις προωθήσει στο εσωτερικό της. Οι κοινέ αξίες, όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, είναι το θεμέλιο της ελευθερίας, ασφάλειας και ευημερίας της Υπήρου μας. Αυτές οι αξίες πρέπει να ε, συνενώνουν τα κράτη-μέλη πρέπει να γεφυρώσουμε τις ε, εσωτερικές διαιρέσεις της Ευρώπης. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμβασμός στην εφαρμογή του κράτους δικαίου. Η Φιλανδία καλωσορίζει θερμά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύνδεση του πολιτού ε, δημοσιονομικού πλαισίου με το κράτος δικαίου. Είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί ένας ε, ισορροπημένος μηχανισμός για να εφαρμοστεί αυτή η αρχή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο πιο σημαντικό ακρογωνιαίο λήθο που καθορίζει τη θέση τη Φιλανδία όσον αφορά την εξέλιξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νομισματική Ένωση είναι ο σεβασμό των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί και να υπάρξει ε, αποτελεσματική εφαρμογή τους. Στηρίζουμε ισχυρά μια Ευρώπη που επιτυγχάνει αξιοπιστία μέσω συγκεκριμένης δράσης. Το 2015 η κυβέρνησή μου ανέλαβε ενώ είχαμε ένα δημόσιο έλλειμμα περίπου 3,5% σε σχέση με το ΑΕΠ. Το κατεβάσαμε στο 2% μέσω ε, εποδίνων ε, εξοικονομήσεων σε σχέση με το ΑΕΠ πάντα το 2%. Βελτιώσαμε τα δημοσιονομικά μέσω μεταρρύθμισης ε, των συντάξεων και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και άλλων κοινωνικών μέτρων. Η εσωτερική υποτίμηση το 4% έγινε μέσω προώθησης της ε, απασχόλησης και της ανάπτυξης. Συμφωνήσαμε με τα συνδικάτα για πάγωμα των μισθών και για περικοπές. Επεκτείναμε κατά 24 ώρες ε, τον ετήσιο χρόνο εργασίας και μειώσαμε τις εισφορές των εργοδοτών στη κοινωνική πρόνοια. Αυτές είναι μόνο ε, κάποιες από τι πρωτοβουλίες μα. Μπορείτε να καταλάβετε, αυτές μας οι ενέργειες δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ωστόσο τώρα, μετά από τρία χρόνια, δεν έχουμε πλέον δημόσιο έλλειμμα. Ο προπολογισμό είναι ισοσκελισμένο και η απασχόλησή μας είναι η υψηλότερη εδώ και 30 χρόνια. Οπότε, η ιδέα ότι πρέπει να λύνονται αυτά τα προβλήματα μέσω μονίμων δημοσιονομικών μεταφορών είναι απαράδεκτη για μας. Η καλύτερη εγγύηση κατά των οικονομικών σοκ είναι ισοσκελισμένοι προπολογισμοί και χαμηλό χρέος. Πολλές φορές τα χρόνια αυτά θυμάμαι αυτό που είπε ο Ζαν Κλοντ Juncker. Όλοι ξέρουμε τι να κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς να επανεκλεγούμε αφού θα το έχουμε κάνει. Εγώ ε, θα ελέγξω στην πράξη αυτό στις ε, περχόμενες εκλογές τον Απρίλιο. Για να δούμε. Τι εννοώ. Παρά τον κίνδυνο, τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις. Η αποτελεσματική εφαρμογή είναι η μακράν καλύτερη μέθοδος για να αποκριθούμε στις ε, σημερινέ και μελλοντικέ προκλήσει. Θέλουμε εφαρμογή τη ενιαία αγορά και πολιτικών για την έρευνα, ανάπτυξη και την καινοτομία. Θέλουμε εφαρμογή των ε, πολιτικών εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Θέλουμε εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών και εφαρμογή των πολιτικών για την καταπολέμηση κλιματική αλλαγή. Η καλύτερη εφαρμογή είναι ο καλύτερο τρόπο για να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή λαϊκισμού και για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, η Φιλανδία θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Θα αναφέρω λοιπόν κάποια σημεία που θα μας απασχολήσουν στην Προεδρία μας. Είναι επίσης θέματα στα οποία θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστεί στενότερα και να κάνει και τα όσα λέει. Θα ξεκινήσω από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το βασικό εργαλείο εφαρμογής της πολιτικής. Κατά την άποψη της ε, Φιλανδίας, το συνολικό επίπεδο του ΠΔΠ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τωρινό ποσοστό. Πρέπει να εστιάσουμε στους τομείς όπου έχει τις καλύτερες δυνατότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετανάστευση, ασφάλεια, ενιαία άγορα, καινοτομία, ψηφιοποίηση και κλίμα. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη να υπάρξει μια ανακατανομή των κονδυλίων της αγροτικής ανάπτυξης εντό του προπολογισμού. Η κοινή αγροτική πολιτική μας δίνει την δυνατότητα να δώσουμε ασφαλή και προσιτά τρόφιμα στους πολίτες και να μπορούν βεβαίως να ζήσουν από τη δουλειά τους και οι αγρότες. Ταυτόχρονα η πολιτική συνοχή ε, δημιουργεί πιο ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ κρατών μελών και εντό των κρατών μελών. Είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των παραδοσιακών πολιτικών τη Ένωση και των νέων προκλήσεων. Είμαι επίση πεπισμένο ότι μπορεί αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Φιλανδία. Δεύτερον, χρειάζεται μια μεταναστευτική πολιτική με μια συνολική προσέγγιση. Πρώτα, οι αιτίε της μετανάστευσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά. Πέρα από την αναπτυξιακή συνεργασία και ανθρωπιστική βοήθεια απαιτούνται το εμπόριο και οι επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να γίνει πιο αποτελεσματική πολιτική των επιστροφών. Η εσωτερική πτυχή της μετανάστευσης είναι στα χέρια μας. Πρέπει να διαχειριστούμε την ε, μετανάστευση μέσω άμεσων μετεγκαταστάσεων από τα στρατόπεδα προσφύγων. Αυτό θα σημάνει μικρότερη πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και λιγότερη λαθρέα διακίνηση. Ταυτόχρονα, η διαχείριση των εξωτερικών σύνορων μας θα πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης, Υπάρχει ανάγκη να προχωρήσουμε με τα πιο πολύπλοκα πολιτικά ζητήματα, όπως ένας μηχανισμός αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια των κρίσεων. Πρέπει να το συμφωνήσουμε αυτό εκ των προτέρων και όχι εν το μέσο μιας κρίσης όπως κάναμε το 2015. Τρίτον, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια που είναι επίσης σημαντική και πρέπει να ενταθεί η Φιλανδία ζητά ενεργά μια φιλόδοξη πρόοδο σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας μαζί με τη Γαλλία. Είναι καλοδεχούμενη λοιπόν αυτή η πρόοδος. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου και της ε, ΠΕΣΚΟ επίσης είναι βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή και στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει ενισχύσει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών στο Ελσίνκι συνεισφέρει στην ετοιμότητα των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις 19 χώρες που συμμετέχουν 16 από τις οποίες είναι κράτη-μέλη της Ένωσης για την ε, προσήλωσή τους ε, σε αυτό. Επίσης, ε, καλώς ορίζω και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη αν θέλουν να ενταχθούν. Τέταρτον, πρέπει να βελτιωθεί η ενιαία αγορά. Είμαστε η καλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο. Πέρα από τις καινοτομίες και το εμπόριο, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας θέσεων εργασίας. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ειδικά στις υπηρεσίες και τα ψηφιακά προϊόντα. Η βελτίωση της κατάστασης εξαρτάται από εμάς. Σας ε, ζητώ λοιπόν να καταλήξετε σε μια κοινή αντίληψη για να περάσουν οι 35 προτάσεις που είναι ακόμα αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Κοιτώντας προς το μέλλον, ελπίζω η νέα Κομισιόν να έχει μια πιο γενική προσέγγιση όπου θα συνδέονται καλύτερα η ενιαία αγορά, η ψηφιοποίηση, η βιομηχανική πολιτική και η ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ανάπτυξη που θα κοιτάει προ το μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κινητικότητα δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη και άλλα. Επίσης, πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα εφαρμόζοντας τις αρχές του κοινωνικού πυλώνα. Παραδείγματο χάρη έχει μεγάλη σημασία να προωθηθεί η ισότητα στον χώρο εργασίας και να ενισχυθεί το επίπεδο εκπαίδευση όλων των πολιτών. Πέμπτον, η εμπορική πολιτική έχει μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νέες θέσης εργασίας. Όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, είμαι ικανοποιημένος από τα τελευταία επιτεύγματα που είχαμε, τη σύναψη συμφωνιών με Ιαπωνία, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, Μεξικό και Καναδά. Και εύχομαι να ολοκληρωθούν ε, σύντομα οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Όμως, είναι επιβλαβές εάν οι μεγάλοι παίκτες συνεχίζουν να υψώνουν εμπορικά τείχη, τα οποία πρέπει να ρίξουμε ειδικά από την σκοπιά των μικρότερων χωρών ε, η ζημιά μπορεί να είναι μοιραία. Πρέπει να σεβόμαστε τους κοινού κανόνες του εμπορίου. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή. Η έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή μας υπενθύμισε και πάλι πως ε, πλέον απειλείται η ζωή στη γη. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα συμπεράσματα της επιστήμης. Ε, πέρα από τις απειλές βλέπω πάρα πολλές ευκαιρίες. Ως μηχανικός σκέφτομαι και προσανατολίζομαι προς λύσεις και προς την τεχνολογία. Είμαι σίγουρος πως ε, καθώς ο κόσμος προχωρά προς ανάπτυξη με χαμηλό άνθρακα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, φιλόδοξης κλιματικής πολιτικής και έτσι θα έχουμε και νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Πρέπει να ληφθούν μέτρα σε τρία μέτωπα. Εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα και ε, απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα και νέες τεχνολογίες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την ε, σκανδιναβική συνάντηση για το κλίμα στο Ελσίνκι και οι σκανδιναβικές χώρες υποσχέθηκαν να αυξήσουν το επίπεδο φιλοδοξίας μέχρι το 2020. Θέλουμε να παίξουμε έναν καταλητικό ρόλο για να περιοριστεί η παγκόσμια θέρμανση στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Επίσης, κατά τη διάρκεια συζητήσεων στο Κοινοβούλιο της Φιλανδίας, 8 κόμματα της χώρας έθεσαν τον στόχο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα πριν το 2050. Αυτό απαιτεί αυστηροποίηση των υποχρεώσεων ε, που έχουμε για το 2030 στο 55% τουλάχιστον του επίπεδου 1990. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπομπών είναι το πιο οικονομικό και αποτελεσματικό σύστημα για την ε, μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα έχει δημιουργήσει το σύστημα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να καθοδηγεί τους ε, παραγωγούς προς τη μείωση των ε, εκπομπών κατά τρόπο αποτελεσματικό. Έχουμε προτείνει, έχουμε πει ότι νέοι τομείς, ε, η ψήξη και η θέρμανση δηλαδή των κτηρίων πρέπει να περιληφθούν στο σύστημα ITS, το σύστημα των ανταλλαγών. Επίσης, ε, πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς μια κυκλική και βίο οικονομική δραστηριότητα. Ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα δράση για τη βιοοικονομία πρέπει άνευ καθυστερήσεως να υλοποιηθεί. Μια μικρή λεπτομέρεια. Η κυβέρνησή μου αποφάσισε να μην ε, ετοιμάσει δωράκια της Προεδρίας, αλλά να κάνει τη σχετική εξοικονόμηση από τους ε, πόρους σε άνθρακα που θα προξενούσαν τα ταξίδια τα αεροπορικά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Επίσης, πρέπει να μιλήσουμε για τις ε, δεξαμενές άνθρακα. Καταβόθρες άνθρακα. Έχουμε 4 εκατομμύρια εκτάρια δασών και 5 ε, δισεκατομμύρια εκτάρια δασών και 5 δισεκατομμύρια εκτάρια ε, καλλιεργήσιμης γης. Με ξαφνιάζει λοιπόν το πόσο πολλοί άνθρακα θα μπορούσαμε να συγκρατήσουμε από τα χωράφια εάν κάναμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα καλλιεργούμε. 100 ε, γεωργοί άνθρακα, ανθρακογεωργοί θα μπορούσαμε να τους πούμε, μπορούν να δοκιμάσουν τώρα τις νέες αυτές πρακτικές στη γεωργία και μπορούμε να, να κάνουμε αντίστοιχους σχεδιασμούς και για τα δάση. Μόνο η Αφρική ε, χάνει 2 εκατομμύρια εκτάρια δασών κάθε χρόνο όσο είναι δηλαδή ολόκληρη η έκταση της Σλοβενίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων μας λέει στην έκθεση για, τα παγκόσμια, για την κατάσταση των δασών στον κόσμο ότι πρέπει να ε, εστιαστούμε περισσότερο στα δάση αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Ένα συγκεκριμένο βήμα θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε την εξωτερική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση των συνολικών ε, καταβοθρών ε, ή δεξαμενών άνθρακα. Έχει προτείνει λοιπόν ένα, ένα ευρωπαϊκό ε, ταμείο για τα δάση της Αφρικής η Φινλανδία με αντίστοιχες επενδύσεις που θα είχαν σημαντικές σημαντικό αντίκτυπο για, τα, για το κλίμα αλλά και για τις γεωργικές θέσεις εργασίας. Ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε το τεχνικό δυναμικό για να συγκρατούμε περισσότερο άνθρακα, διοξίδιο του άνθρακα από τον αέρα και να το μετατρέπουμε σε άλλα προϊόντα. Έχουμε τεράστιο δυναμικό έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομία στον τομέα αυτό. Επίσης πρέπει να στραφούμε με καινοτόμους τρόπους για να αναζητήσουμε νέες, ε, νέα κίνητρα και νέες μεθόδους με εφαρμογές στην αγορά που θα εξασφαλίσουν την αύξηση των δεξαμένων άνθρακα. Το κύριο μήνυμα που θέλω να απευθύνω είναι ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και πρέπει να τα κάνουμε ταχύτερα. Πρέπει να μειώσουμε εκπομπέ, πρέπει να ενισχύσουμε τι ε, καταπόθεση άνθρακα και να υιοθετήσουμε νέε τεχνολογίε για τη συγκράτηση του οξυδίου του άνθρακα από τον ατμοσφαιρικό αέρα ή, αμε, ίσω και αμέσω από, την από πηγή τη εκπομπή. Αγαπητοί Ευρωπαίοι συμπατριώτες, Αμέσως μετά τι ε, ευρωεκλογέ, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει συμφωνία για το φιλόδοξο και πλήρες ε, σχέδιο που ονομάζεται ε, θεματολόγιο για τη στρατηγική. Πέραν των θεμάτων του κλίματος θα πρέπει να σταθούμε και στην ανάπτυξη και την ασφάλεια. Βεβαίως και τα θέματα του κράτους δικαίου παραμένουν κρίσιμη σημασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν και απευθύνω μία έκκληση για πιο συγκεκριμένες δράσεις ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση με ουσιαστική υλοποίηση του δικαίου και με περισσότερες ευθύνες. Ευθύνες που σημαίνει και εγώ αναλαμβάνω ευθύνη για τον εαυτό μου, αλλά αναλαμβάνω ευθύνη και για τους γύρω μου και για το περιβάλλον μου και άρα και για ολόκληρο τον ε, πλανήτη όπως και για την οικονομία. Α ε, θυμόμαστε ότι εμεί έχουμε εδώ ως ρόλο να διαφυλάξουμε ένα καλύτερο μέλο για τους νέους μας και για τις επόμενες γενιές. Για το δικό τους το καλό. Για το μέλλον απαιτείται να έχουμε μια αποφασισμένη, αποφασιστική, αποτελεσματική και ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως απαραίτητο είναι να επιδείξουμε έργο δεν μπορώ παρά να τονίσω αυτή τη σημασία και γι' αυτό τη λέξη implementation, εφαρμογή, υλοποίηση, την έχω επαναλάβει τόσες φορές μέσα στην ομιλία μου. Οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης θα ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, λαμβάνοντας αποφάσεις και υλοποιώντα. τες, τόσο στο εσωτερικό τους όσο και εδώ στι Βρυξέλλες. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον ε, Πρωθυπουργό Σιπηλά για την ομιλία του οποίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρακαλώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Ζων Κλοντιουνκέ, να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και ο Γύρκη, κατά έναν και εγώ, με μεγάλη χαρά συναντούμε τον φίλο Πρωθυπουργό της Φινλανδίας. Η Φινλανδία το 1995 κατέστη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατατύχει την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα ανέλαβα εγώ καθήκοντα ως Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Από τότε μέχρι σήμερα, ε, πότε, πότε δουλεύει η Ευρώπη ικανοποιητικά. Και σημείωσα εξ αρχής, διαπίστωσα εξ αρχής, ότι από την πρώτη μέρα της ένταξής της η Φινλανδία είχε στάσει και συμπεριφορά σαν να ήταν ιδρυτικό μέλος, σαν να ήταν ανέκαθεν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλω να πω ότι ορισμένα από τα ιδρυτικά μέλη θα μπορούσαν πολλά να αποκομίσουν αν ακολουθούσαν το παράδειγμα της Φιλανδίας και ακολουθούσαν αυτή τη συμπεριφορά. Η Φιλανδία από την ε, ένταξή της έδειξε πάντα μία τάση να αφουγκράζεται οι κυβερνήσεις της όλες ήξεραν να τίνουν ευικονούς η Φινλανδία αφού γκράζεται, αντιλαμβάνεται αυτό που ακούει και μετατρέπει σε πράξη αυτό που έχει αντιληφθεί στην πολιτική. Έχοντας ξεκινήσει με τον Πάβο Λίπον ως Πρωθυπουργό, με τον Κατάινεν μετά, με σένα εδώ, να, αργότερα, πάλι τρεις Πρωθυπουργούς σήμερα, από την Φιλανδική Προεδρία, ε, Φιλανδική ημέρα σήμερα, σπάνιο μεν, αλλά χρήσιμο Τρεις Φιλανδοί θα περάσουν από την ε, Επιτροπή σήμερα. Και έχουμε λοιπόν και την επόμενη Φιλανδική Προεδρία στον ορίζοντα, μια Προεδρία με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, καθώς ξεκινάει η Προεδρία της Φιλανδίας μετά τις ευρωεκλογέ. πριν από, την, από τον διορισμό του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής και της Επιτροπής Λογικά και του νέου διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Επομένως, αναλαμβάνεται καθήκοντα ως Προεδρία σε μια περίοδο που χρειάζεται πολύ επιδεξιότητα στη διαχείριση των Ευρωπαϊκών και της ε, Προεδρίας, όπως άλλωστε έχει αποδείξει η Φιλανδία ότι μπορεί να πράξει. Το έχει αποδείξει και σε προηγούμενες ε, Προεδρίες της. Όσον αφορά τη σχέση Φιλανδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι καλύτερες δεν θα μπορούσαν να είναι. Έχουμε σχέση απόλυτη εμπιστοσύνη στη συνεργασία μα, όπω άλλωστε είδαμε και κατά την εγκαθίδρυση του μηχανισμού ασφάλεια και άμυνα, όπω άλλωστε συμβαίνει και στον τομέα τη ενέργεια και των κλιματικών αλλαγών, όπω άλλωστε συμβαίνει και στην ανάπτυξη των υποδομών ε, διασυνδεσιμότητας στην υπεθροτή ε, της και εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα χάρη στην ε, ευκαιρία που μας δίνει η ανάληψη της Προεδρίας από την Φιλανδία να αναπτυχθεί περισσότερο η διάσταση του ε, βόρειου αρκτικού κύκλου. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ε, μια περιοχή στο Βόρειο βορειοαρκτικό κύκλο που παρουσιάζεται διπλάσια αύξηση θερμοκρασίας από ό,τι στην υπόλοιπη Ιφίλιο και άρα πρέπει να, υπάρχει, να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, άλλωστε υπάρχει και σχετικό συμβούλιο. Τον Νοέμβριο που ήρθα στη Φινλανδία, συζήτησα με τον ε, Πρωθυπουργό την ιδέα για μια σύνοδο κορυφής των χωρών του Βόρειου Αρκτικού Κύκλου, διότι θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η περιοχή αυτή, ο Βόρειος Αρκτικός, να μπει ως κύρια προτεραιότητα στην, ε, στο θεματολόγιο των ευρωπαϊκών εργασιών. Ταυτόχρονα όμως έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία πράγματα η Φινλανδία και ως Προεδρία και μπορεί να κάνει και αυτό ελπίζω να συμβεί με την εμβάθυνση και της Νομισματικής Ένωσης κατά τη διάρκεια της ε, Φινλανδικής Προεδρίας, με την Τραπεζική Ένωση, με την ολοκλήρωση της κεφαλαϊκής αγοράς που μπορεί να μας εξασφαλίσει η Φιλανδική Προεδρία. Υπό τη Φιλανδική Προεδρία πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε και, αυτό είναι στο επίκεντρο αυτής της, αυτού του προγραμματισμού, και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτή είναι η μεγάλη δουλειά, η σκληρή δουλειά που έχει μπροστά της Φιλανδική Προεδρία, στην οποία πιστεύω ότι μπορεί να στηριχθεί απολύτως στην ε, βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οτιδήποτε χρειάζεστε θα το προσφέρουμε έτσι ώστε στο Συμβούλιο το ευρωπαϊκό του Οκτωβρίου να ολοκληρωθεί αυτό το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει εφέτος να ολοκληρωθεί, να κλείσει δηλαδή ως συμφωνία. Ιδάλλως χάνουμε πολλές ευκαιρίες για κατάθεση προτάσεων προγραμμάτων και χρηματοδότησή τους. Θα ήμουν επίσης ευγνώμων προς τη Φιλανδική Προεδρία και μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά και στον τομέα τη εμβάθυνση Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θα παρακαλούσα να ε, εισακούσει τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των διαθροτικών μέσων και τη σταθεροποίηση τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης αλλά και τη ανταγωνιστικότητά τη και τη ε, στεναρότητά τη έναντι εξωτερικών κλειδονισμών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μα. Έχουμε ένα ζήτημα για το οποίο ο πολίτης περιμένει να έχει τη δυνατότητα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να είναι σε θέση να αντιδράσει καλύτερα στην επόμενη κρίση που θα βρούμε μπροστά μας. Και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τη Φιλανδική Προεδρία, προ την Φιλανδική Κυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι σκοπεύει να αποδώσει μεγάλη σημασία στο επενδυτικό σχέδιο του Γύρκη και το δικό μου. Ε, έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη ξεκινήσει με την υλοποίηση περί τα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Φινλανδία. Ελπίζω να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και σας εύχομαι κάθε επιτυχία τον Απρίλιο, κάθε επιτυχία για την ανάληψη της Φιλανδικής Προεδρίας στη συνέχεια. Κάθε επιτυχία για το μέλλον. Ευχαριστώ. Θα ήθελε άλλος βουλευτής να εγγραφεί στο κατάλογο για τη διαδικασία Catch the Παρακαλώ, εάν ναι, παρακαλώ να το πράξετε αμέσως. Ιδάλλως θα κλείσω τον κατάλογο της ηλεκτρονικής εγγραφή, την ηλεκτρονική εγγραφή στον κατάλογο και παρακαλώ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της ε, ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κύριο Μάνφρετ Βέμπερ, να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι μια κρίσιμη συγκυρία όπου τον Απρίλιο θα εκφραστεί ο λαός σας και η ευρωπαϊκή λαή τον Μάιο. Θα έχουμε δημοκρατικές λοιπόν εκλογές τους επόμενους μήνες. Ξέρετε ότι η πρωτεύουσά σας, ε, το Ελσίνκι, είναι για εμένα και για το κόμμα μας ε, ζωτική σημασία. Εκεί πήρα το χρήσμα του υποψηφίου στο συνέδριό μας. Και αυτό ακριβώς αναμένουν οι πολίτες να έχουμε συζητήσεις, να υπάρχουν υποψηφιότητες και μετά θα επιλέξουν οι πολίτες για το μέλλον μας και την κατεύθυνση της πορείας μας. Αυτές είναι οι αρχές της εθνικής και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Θα είναι στο κέντρο των εξελίξεων των επομένων μηνών. Θέλω να συμμεριστώ μερικά σημεία τα οποία αναφέρατε. Να σα συμμεριστώ τις γνώση, τις σκέψεις μου δηλαδή. Στηρίζουμε αυτά που λέτε για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μπορεί να φαίνεται τεχνικό αυτό το θέμα, μπορεί να έχει να κάνει με τι αγορέ, μπορεί να φαίνεται τεχνοκρατικό και ότι αφορά μόνο τι επιχειρήσει. Όχι. Είναι το μέλλον των παιδιών μα. Είναι θέμα βιαισιμότητα. όταν αναφερόμαστε στην δημοσιονομική πειθαρχία. Και το ΕΛΚ και σε εθνικό επίπεδο με τον κύριο Όρπα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με εμά και ο Γύρκη βεβαίω, κατά είναι, είναι στο πλευρό σα. Θα μα έχετε πάντα στο πλευρό σα αν θέλετε να επιδιώξετε αυτήν τη βιωσιμότητα. Γιατί η βιωσιμότητα σημαίνει μέλλον. Δεύτερον, αντιδρώντα στην ε, ομιλία σα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, εδώ θα σα επικρίνω κάπω. Γιατί ξεκινήσατε την ε, αναφορά σα στο πολιτέ πλαίσιο λέγοντα ότι πρέπει να καθοριστεί το ποσό. Αυτό μα λένε πάντα οι εθνικοί ηγέτες Νομίζω πω δεν είναι σωστή προσέγγιση αυτή. Η σωστή προσέγγιση είναι ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι τα καθήκοντά μα. ε, τι απαιτήσει υπάρχουν έναντι τη Ένωση. Πολλοί ηγέτε λένε πρέπει να καθορίσουμε του πόρου, αλλά μετά θέλουμε ισχυρού ελέγχου στα σύνορα, θέλουμε κυβερνοασφάλεια, θέλουμε περισσότερη καινοτομία στην Ένωση. Αν αυτέ είναι απαιτήσει έναντι τη Ευρώπη, τότε τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν σωστά. Πρέπει να συμβάλλουν στον προπολογισμό. Πρέπει να υπάρξει επαρκή χρηματοδότηση για να ανταποκριθούμε στι προκλήσει των καιρών. Πρέπει λοιπόν πρώτα να αναφερθούμε στι προκλήσει των καιρών. Το τρίτο σημείο που θα αναφέρω στη σύντομη παρουσίασή μου είναι το πιο δύσκολο για όλου μα. Αυτό μας είπαν και 35.000 παιδιά όταν ε, διαδήλωσαν τις προηγούμενες εβδομάδες στην Ευρώπη. Καλή και ο Πάπας ε, Φραγκίσκος για να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια τη γη. Είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αναφερθήκατε αναλυτικά σε αυτό. Υπογραμμίζω. Ποιε πρέπει να είναι οι αρχέ που εμεί ω ΕΛΚ θεωρούμε ότι πρέπει να κυριαρχήσουν σε αυτή την αντιμετώπιση. Μία αρχή είναι ότι η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή δεν είναι να απαγορεύουμε διάφορε δραστηριότητε και προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν να λέμε στου πολίτε ότι δεν μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο και να πάνε στη Μαγιόρκα για διακοπέ γιατί αυτό αυξάνει το αποτύπωμα άνθρακα. Όχι, δεν είναι η δική μα προσέγγιση. Ελπίζουμε στο μέλλον να πηγαίνουν ε, οι ταξιδιώτε στη Μαγιόρκα με αεροπλάνα που δεν θα μολύνουν. Αυτή είναι η προσέγγιση. Δεν μπορούμε να πούμε στι αναπτυσσόμενε χώρε ή στι αναδυόμενε οικονομίε ότι θα πρέπει να μην αναπτυχθούν περισσότερο. Δεν είναι απάντηση αυτό. Η απάντηση είναι ότι εμεί ω Ευρωπαίοι Πρέπει να του παράσχουμε σε αυτέ τι αναπτυσσόμενε χώρε τι αναγκαίε τεχνολογίε, ούτω ώστε η ανάπτυξή του να μην έχει επίπτωση στο κλίμα. Αυτή είναι η απάντηση. Η καινοτομία είναι η βασική αρχή για μα. Δεύτερο σημείο. Για το διοξείδιο του άνθρακα. Πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτε τι κάνουμε. Οι πολίτε πρέπει να υιοθετήσουν τι αλλαγέ. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πολλοί ανησυχούν για αυτέ τι αλλαγέ. Βλέπετε τι διαδηλώσει των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία και πολλοί και εδώ στην αίθουσα. Μπορούμε να πληρώσουμε υψηλότερε τιμέ ενέργεια, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι συμπολίτε μα. Πρέπει λοιπόν να επέλθουν αυτέ οι αλλαγέ με τέτοιο τρόπο που να τι αποδεχθούν οι πολίτε. Να ενστερνιστούν την άποψή μα. Πρέπει να κερδίζουμε από αυτήν την αλλαγή και όχι να χάνουν κάποιοι. Και τέλο, για την κλιματική αλλαγή του διοξείδου του άνθρακα, μαζί μπορούμε να δράσουμε. Εμεί καταστήσαμε δυνατή τη Συμφωνία των Παρισίων. Εμεί κάναμε τα βήματα για να μειωθούν οι εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα, διοξιδίου του άνθρακα. Εμείς είμαστε πρωτοπορία παγκοσμίω στην καταπολέμηση, στη μείωση δηλαδή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αποκινούμε τους ε, πολίτες μας μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο ομιλητής, Κόφοντ, για τη σοσιαλιστική ομάδα. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ. Η πατρίδα σας συμφωνητές είναι ηγετική δύναμη σε πολλού τομεί στην καθαρή ενέργεια, την ισότητα των φύλων, τα κοινωνικά θέματα. Η Transparency International ε, κατέταξε στην υψηλότερη βαθμίδα διαφάνειας και μη διαφθορά στην Φινλανδία στον κόσμο. Ε, βεβαίως πρέπει να πω ότι μας έχετε προλάβει εμάς σε ορισμένα θέματα όπως είναι η ενέργεια, έστω του Δανούς δηλαδή. Πάντως η, Δανία, η Φινλανδία δείχνει ότι μπορεί μια μικρή χώρα να ε, βρίσκεται μπροστά στον κόσμο, έστω και αν γεωγραφικά είναι πιο απομακρυσμένη. Θα ήθελα όμως ε, να πω ότι δεν είδα σε εσά στην ομιλία σας αυτή τη φιλοδοξία να καταστείτε πρωτεργάτης, να ηγηθείτε, να σπρώξετε την Ευρώπη προς την βιώσιμη ανάπτυξη, την δίκαιη ανάπτυξη, την ε, ανοιχτή σε όλους ανάπτυξη. Πού ήταν τα λόγια που θα λέγανε θα κάνω τη ζωή των Ευρωπαίων καλύτερη. Τα όσα μας είπατε περισσότερο μου θύμισαν τα νεοφιλελεύθερα σλόγγαν της ε, χθεσινής μέρας και όχι τη, τα φιλόδοξα σχέδια για το αύριο. Εμείς ε, οι σοσιαλιστές έχουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την Ευρώπη. Ε, πιστεύουμε ότι η γη μας... η πόροι μας κινδυνεύουν από την ε, ρήπανση, από την κλιματική αλλαγή. Ο ατμοσφαιρικός αέρας που αναπνέουμε, το νερό που πίνουμε, το χώμα πάνω στο οποίο περπατάμε είναι το μέλλον των παιδιών μας και έχουμε καθήκον να τα υπερασπιστούμε. Ωστόσο και οι πολίτες μας και οι εργαζόμενοι έχουν κουραστεί να πληρώνουν αυτό το λογαριασμό ενός πιο βιώσιμου τρόπου αναπαραγωγής και με δυσφορία βλέπουν ότι οι μεγάλες πολυεθνητές ρηπαίνουν χωρίς όμως να πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί σε δίκαιους φόρους. Πρέπει αυτό να αλλάξει πια. Πρέπει να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης να καταστεί ένας, ένα πραγματικό σύμφωνο βιωσιμότητα για την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν και έχουμε εμεί ένα σχέδιο για να προχωρήσουμε πιο με ένα πιο, πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγή για να είναι πιο ε, δίκαιε συνθήκε και η μετάβαση για τον πολίτη και την Ευρώπη. Και σήμερα Καλό τη Φινλανδία να ενώσει τις δυνάμεις της σε αυτό το σημαντικό αγώνα, να έρθει κοντά μας. Πρέπει εμείς να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση όπως εμείς την εννοούμε και όχι να αφήσουμε να επικρατήσουν οι δυνάμεις της καταστροφής. Πρέπει εμείς να ορίσουμε τους κανόνες και τους όρους του παιχνιδιού. Η απληστία ορισμένων ελίτ και ο η ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση μας οδηγούν στην καταστροφή. Μόνο έτσι λοιπόν με την κατάλληλη φορολόγηση, με τις συνθήκες εργασίας για όλους ισότιμες και τον κοινωνικό πυλώνα που δεν άκουσα το κουβέντα να ξοδέψετε για αυτόν που με τόση δυσκολία υιοθετήσαμε εδώ στην Ευρώπη. Κύριε Πρωθυπουργέ, η δίκαιη φορολόγηση είναι το θεμέλιο του κράτους ε, προνοίας της Ευρώπης που είναι άλλωστε μοντέλο το ε, κοινωνικό κράτος στη Βόρεια Ευρώπη, στη Φιλανδία και τις άλλες χώρες. Ε, είδαμε από μία μελέτη την προηγούμενη εβδομάδα από τον καθηγητή Μέρφυ ότι 800 85 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το, το κενό στην χρηματοδότηση που χάνεται, στου σπόρου που χάνεται από την ε, φορολογία που δεν καταβάλλεται από τι μεγάλε πολιεθνικέ. Έχουμε τεράστιο δυναμικό λοιπόν να αντλήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουν οι κατάλογοι με τους παραδείσους φορολογικούς, ε, όχι μόνο έξω από την Ευρώπη αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Γιατί ο πολιτή δεν καταλαβαίνει πώ είναι δυνατόν εμεί οι πολίτε να πληρώνουμε όλο και πιο υψηλού φόρου, όταν η Facebook, η Google και άλλοι μεγάλοι μεγάλη κολοσσή ε, πληρώνουν ελάχιστου ή και καθόλου φόρου στην Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να προστατέψουμε το κράτο προνοία ε, όχι μόνο για να είναι ελεύθερο ο ανταγωνισμό, αλλά και δίκαιο ο ανταγωνισμό, θεμητό ο ανταγωνισμό για όλου αυτού. Πρέπει να διωχθούν και πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν αυτοί οι οποίοι αποφεύγουν την καταβολή φόρου. Η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων και τη ιατροφαρμακή θρησκευτικής ε, πρόνοιας ε, και περίθαλψης κύριε Πρωθυπουργέ δεν θα είχε ε, ίσως ε, πραγματοποιηθεί στη Φινλανδία εάν υπήρχαν οι πόροι αυτοί που έχουν εξεφύγει. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε να μείνει κανείς έξω κύριε Πρωθυπουργέ. Βλέπουμε κάποιες δυνάμεις προσπαθούν να διαλύσουν την Ευρώπη. Χρειάζονται όμως αυτές οι ριζικέ αλλαγέ που θα οδηγήσουν στην κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο αγώνα μα εμά των σοσιαλδημοκρατών τη Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι οι φιλελεύθεροι και οι άλλοι προοδευτικοί θα ενωθούν στον αγώνα αυτό. Ευχαριστώ per il gruppo dei conservatori dei ε, ε, και μεταρρυθμιστέ, ε, τον λόγο έχει η κυρία Ρόχναν Λέρνερ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κοινό μας στόχο είναι σίγουρα να αυξηθεί η ευημερία. Η αύξηση τη Ευρωπαϊκή ευημερία και αυτό θα ήθελα ακριβώς να τονίσω το θέμα της μετανάστευσης, την ασφάλεια των πολιτών, την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την προστασία των πληροφοριοδοτών. Κύριε Πρωθυπουργέ, είχατε δηλώσει δημοσίως το 2015 πως ε, θα θέσετε στην διάθεση ετούν τον άσυλο τη μονοκατοικία σας με τις εννέα κρεβατοκάμαρες. Αλλά αυτό αναπαράχθηκε από τα ΜΜΕ και πολλοί νέοι από το Ιράκ είπαν ότι το άκουσαν αυτό και επέλεξαν ειδικά τη Φιλανδία. Πέρα από αυτό Ε, διάβαζαν ε, τις διάφορες ε, περιγραφές για την δωρεάν παροχή υγείας, εκπαίδευσης, την καθαρή φύση, τις ωραίες γυναίκες που τους περιμένουν, όλα αυτά στο Αλαράμπια που ήταν σαν τα ουρί του παραδείσου. Λοιπόν, εσείς απευθύνατε αυτήν την πρόκληση, έκτοτε έχουμε σεξουαλικά εγκλήματα και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών έχει επιδεινωθεί. Αναγνωρίζετε τώρα ότι η πρόσκλησή σας αυτή οδήγησε στο να έρθουν πολλοί άνθρωποι που τελικά δεν έχουν κάποια βάση για να λάβουν άσυλο. Τα προβλήματα στις χώρες προέλευσης δεν μπορούν να λυθούν με το να μετακινηθεί ο πληθυσμός του στην Ευρώπη. Τα προβλήματα πρέπει να λυθούν εκεί. Δεν μπορεί η Ευρώπη να γίνει το Ταμείο Ενεργείας ε, του πλανήτη. Λοιπόν, ε, συζητάμε επίσης για την φροντίδα των ε, ηλικιωμένων και ιδιαίτερα για μια εταιρεία που προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες. Μια τέτοια εταιρεία εξοικονόμησε πάρα πολύ κόστη με το να παραμελεί τους ε, ασθενείς ε, και πολλοί προσπάθησαν να αποφύγουν τους ε, φόρους και μετέφεραν το κεφάλαιο του σε φορολογικούς παραδείσους. λοιπόν πολλά προβλήματα που εμφανίζονται. Πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν μια κουλτούρα όπου όλα τα εγκλήματα, παραδείγματο χάρη η παραμέληση αυτών των ε, ηλικιωμένων, ε, η φοροαποφυγή και τα περιβαλλοντικά εγκλήματα θα πρέπει να δηλώνονται αμέσως στις αρχές όταν παρατηρεί κανείς ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να θεωρούνται υπέρμαχοι του δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, κάποια κανάλια που θα τους επιτρέπουν να το κάνουν αυτό με τρόπο εύκολο και ανώνυμο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη Φιλανδία. Τον λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, ο κύριος Φερχοφστάτ. Κύριε Πρωθυπουργέ, και εγώ ξεκίνησα ως Πρωθυπουργό Ζων Κλοντ Κέρ, στη Φινλανδία, θα θυμάσαι ίσως. Η πρώτη σύνοδο κορυφή στην οποία έλαβα μέρο ως Πρωθυπουργό ήταν το Τάμπερε. Να, 98, τα θυμάμαι πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα ότι είχαμε στάρανδο στο μενού στη Σύνοδο. Και επίση ότι εκεί αποφασίστηκε μια κοινή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ακόμα αγωνιζόμαστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη για το σκοπό αυτόν. Χάρηκα από τα όσα είπατε, γιατί ξεκινήσατε στην ομιλία σας με τον Άκιο και έχω κι εγώ μια παράθεση των λόγων του, με βοήθησε ο Νίλς βέβαια, ο συμπατριώτη σας, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τις ιδέες της κοινωνίας των εθνών και να χτίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του 20 τα είπε αυτά. Ένα εγχείρημα υπέροχο, ένα εγχείρημα που πρέπει να οικοδομηθεί και βεβαίως στην ε, παρέμβαση σας άκουσα τρία σημαντικά θέματα στα οποία θέλω να σταθώ. Καταρχάς, Ευρωζώνη και διακυβέρνησή της και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν χρειάζεται μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, δεν χρειάζεται δηλαδή να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση για να αντικατασταθεί η δουλειά που δεν κάνουν στο ιστορικό τα κράτη-μέλη από την εισαγωγή νέων μέτρων. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει, να κάνουν τη δουλειά που έχουν να κάνουν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νέο νόμισμα βεβαίω, το οποίο όμω χρειάζεται και την δημοσιονομική δυνατότητα με τα ε, ασφαλή στοιχεία ενεργητικού σε παγκόσμιο, με παγκόσμια απήχηση που θα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο που θα αποτελεί ταυτόχρονα όμως και την ασφάλειά μας έναντι των λεγόμενων ασυμμετρικών ε, κλειδονισμών. Γιατί αυτό δεν μπορούν μόνο τους τα κρατη το καθένα να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή συμφωνώ μαζί σας μεν, αλλά το ένα συμπέρασμα αντιφάσει και με το άλλο. Και το δεύτερο, εσωτερική αγορά. Λέτε ότι έχουμε την καλύτερη εσωτερική αγορά του κόσμου. Να το διορθώσω λίγο. Θα μπορούσαμε, ίσως, να είχαμε την καλύτερη εσωτερική αγορά του κόσμου. Εάν είχαμε μια ενιαία αγορά και στους τομείς της ψηφιακής αγοράς, των κεφαλαίων, της ενέργειας. Και σε αυτό χρειάζεται ένας ρυθμιστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άπαξ και υπάρξει αυτό, αυτομάτως θα δούμε να αναδύεται η εσωτερική αγορά, η ενιαία αγορά για τα ψηφιακά, για τα κεφάλαια, για την ενέργεια. Η άμυνα, τρίτη παρατήρηση η μεγαλύτερη διασπάθηση κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται αυτή τη στιγμή στο ότι δεν υπάρχει μια γνήσια ευρωπαϊκή άμυνα. Δαπανούμε χρήματα και για την άμυνα των... Ε, χρήματα περισσότερα από ό,τι οι Αμερικανοί, ακόμα και οι Ρώσοι, αλλά δεν έχουμε την αμυντική δυνατότητα. Γιατί, γιατί επαναλαμβάνουμε τέτοια πράγματα επί 28 και ελπίζω ότι θα καταστεί η Ένωση Αμυντική προτεραιότητα της Φιλανδικής Προεδρίας. Τώρα η συμπρόεδρος... Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ που ήρθατε στη συζήτηση αυτή για το μέλλον της Ευρώπης. Στιγμή αυτή που μιλάμε, 10.000 ε, μαθητές που κάνουν πορεία στους δρόμους ε, εδώ πέρα και στη Φιλανδία και μας δείχνουν πραγματικά ότι πρέπει οι άνθρωποι και ο πλανήτης ε, να προηγηθούν ε, των κερδών. Λοιπόν, σας παρακαλώ να δεσμευτείτε για το μέλλον, να ακούσετε τους νέους και να επενδύσετε στο μέλλον όταν μιλάμε για την προστασία του κλίματος, την εκπαίδευση και την συνεργασία των Ευρωπαίων. Στην προστασία του κλίματος η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τεράστια ευθύνη και κάθε κράτος μέλος πρέπει να παίξει τον ρόλο του. Και χαίρομαι που αναφέρατε το ότι είστε προσιλωμένο σε αυτό, θέλετε να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Ωραία πράγματα και αναφέρατε και την σημασία των καταβοθρών διοξιδίου του άνθρακα και η Φιλανδία βεβαίως είναι ευτυχής που έχει κάτι τέτοιο τα ωραιότατα φιλανδικά δάση και κυρίως χάρη στα δάση της η Φιλανδία έχει γίνει το κράτος πρόνοιας που είναι σήμερα αλλά υπάρχει και ένα σημαντικός παράγοντας στην κλιματική πολιτική εχμαλωτίζουν το ισοδύναμο 20 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. Οπότε είναι προς το κοινό συμφέρον μας να τα διαχειριστούμε με αηφόρο τρόπο. Αλλά σε αντίθεση με τα όσα μας λέτε εδώ πέρα, η κυβέρνησή σας προγραμματίζει υλοτομία στα δάση αυτά, η οποία δεν είναι αηφόρος και είναι ιδιαίτερος υπερβολική. Και έτσι κινδυνεύει αυτός ο πλούτος που έχετε. Ελπίζω λοιπόν μετά την πολύ ωραία σας ομιλία σήμερα η κυβέρνησή σας να αναστρέψει αυτήν την ε, θέση της ε, για να διατηρήσει την κληρονομιά σας και τον ρόλο της ως καταβόθρας διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί εάν είναι να έχουμε μια οικονομία ουδέτερη ω προ το διοξίδιο του άνθρακα, χρειαζόμαστε περισσότερα δάση. Αντί να λέμε στου άλλου να έχουν περισσότερα δάση, πρέπει να διατηρήσουμε τα δικά μα. Χαίρομαι λοιπόν που αναφέρατε ότι θέλετε πιο φιλόδοξους στόχους. Είμαστε στο πλευρό σας. Και χαίρομαι που το κάνετε αυτό και στο Σκανδιναβικό Συμβούλιο. Ε, φέρετε το όμως και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους άλλους πρωθυπουργούς, για να προχωρήσει στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι αποτελεσματική εφαρμογή και οι νέοι, τους οποίους ανέφερα, αυτοί θα διευθύνουν τις χώρες μας, ε, τις ε, κοινωνίες, την οικονομία προσεχώς και ελπίζω πολύ σύντομα. Και πρέπει να τους προετοιμάσουμε γι' αυτό και η Φιλανδία είναι διάσημη για το εκπαιδευτικό τους ε, σύστημα. Όλοι ήρθαν στη Φιλανδία για να αντιγράψουν ε, τα φιλανδικά σχολεία, αλλά λυπούμε για το ότι η κυβέρνησή σας ε, πλέον κόβει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκπαίδευση και την έρευνα. Χρειάζεται περισσότερη επένδυση σε αυτούς το μισό και λιγότερη. Και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε όταν μιλάμε για το ΠΔΠ στο ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή και να συνεισφέρει στην ευημερία όλων των πολιτών και όχι μόνο σε όσων έχουν τα μέσα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχει πολύ περισσότερα καθήκοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα χρειάζεται και επαρκείς πόρους. Δεν θα δεχτούμε λοιπόν μείωση του προϋπολογισμού. Μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τα όσα έχει αναλάβει. Επίση, αναφέρατε πόσο σημαντικές είναι οι κοινέ αξίες, το κράτο δικαίου και η ΕΕ και αναφέρατε τον κίνδυνο του λαϊκισμού και συμφωνώ. Όμως και εσείς συνεργάζεστε με δεξιούς λαϊκιστές, κάποιους από τους οποίους μόλις ακούσαμε, οπότε νομίζω ότι γνωρίζετε πλήρως τις ε, κοινέ προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει η Ήπειρός μας. Ε, εθνικιστικά και ακροδεξιά κινήματα κερδίζουν στήριξη στην Ευρώπη μέσω παραπληροφόρησης. Στις, καλά είναι λοιπόν τα λόγια, αλλά οι πράξεις έχουν σημασία. Εκεί πέρα δείχνουμε ότι είμαστε σοβαροί, ότι θέλουμε ακριβώς να οικοδομήσουμε αυτό το καλύτερο μέλλον μαζί. Καθώς λοιπόν θα έχουμε τη Φιλανδική Προεδρία αυτό το καλοκαίρι, ελπίζω η χώρα σας μετά να είναι στην προοδευτική πλευρά, να μας οδηγήσει προς τα ευρώς για μια ενωμένη και δίκαιη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ για την GUE NGL, τον λόγο έχει ο κύριος Ηλικιώτης. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλωσορίζω από μέρους της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, της Βόρειας Πράσης Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο συζητάμε σήμερα για ακόμα μια φορά το μέλλον της Ένωσης. Ένα μέλλον που καθορίζεται όμως από τη συνέχιση των ίδιων αδιέξοδων και αντιλαϊκών πολιτικών. Των πολιτικών εκείνων που προωθούν τη φτωχοποίηση, τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, προκαλούν την καταστροφή του περιβάλλοντος, προωθούν τη στρατηγικοποίηση, αλλά και το φλερτ των κυρίαρχων πολιτικών κύκλων με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Πόσο πιο δυνατά χρειάζεται να το πούν οι λαοί τη Ένωση πω χρειάζεται ρήξη με τι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ λιτότητα ρήξη με τι πολιτικέ σε βάρο του περιβάλλοντο ρήξη με τι πολιτικέ του κοινωνικού κράτου. μόλι την προηγούμενη εβδομάδα ξεχύθηκα στου δρόμου του Βρυξελό δεκάδε χιλιάδε μαθητέ και εργαζόμενοι για αλλαγή τη πορεία των πολιτικών για το κλίμα. στη γαλλία και αλλού οι εργαζόμενοι εκφράζουν το θυμό και την αγανάκτησή του για τι πολιτικέ οι οποίε του στοχοποιούν. ακόμα και στη φιλανδία που αποτέλεσε παράδειγμα κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης η κοινωνία παρακολουθεί παγωμένη σκάνδαλα που ήταν αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων και της απορρίθμισης στον τομέα της υγείας υποστελέχωση στις στέγες ηλικιωμένων λόγω ιδιωτικοποιήσεων ακατάλληλα φάρμακα στους ηλικιωμένους η αύξηση του κέρδους των εταιριών φροντίδας. πριν από δύο χρόνια από αυτό εδώ το βήμα ο πρόεδρος Γιούνκερ αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει τον κοινωνικό της χαρακτήρα και κινδυνεύει να γίνει η άγρια δύση του κοινωνικού τάμπικ. Δεν παραδέχθηκε όμως ποιε πολιτικές οδήγησαν εδώ. Οι πολιτικές που παράγουν την νεανική ανεργία, τη φτώχεια, τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, ενώ ταυτόχρονα λιένεται το έδαφος για την άνοδο της ακροδεξιάς, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας Όσοι δεν αναγνωρίζουν την αιτία, προφανώς θα συνεχίσουν με τις ίδιες συνταγές και στον ίδιο δρόμο. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη είναι κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική αλληλεγγύη. Χρειάζεται να ανακατανέμεται ο ε, δίκαια ο παραγόμενο πλούτο για κοινωνική δικαιοσύνη, όχι για τι τράπεζε και τι πολυεθνικέ. Ένα άλλο δρόμο ανάπτυξη που να δημιουργεί μόνιμε αξιοπρεπεί θέσει εργασία και πλήρη εργασιακά δικαιώματα να προασπίζεται το δημόσιο χαρακτήρα των στρατηγικών τομέων και υπηρεσιών κάθε χώρα να ενισχύει την κοινωνική προστασία για του αδύναμου και όχι να διανέμει ευχολόγια χωρί μια δεσμευτική ισχύ όπω είναι ο περιβόητο ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα. Ούτε να δίνει πακτολό χρημάτων στο Ταμείο για την Άμυνα ενώ αποκόπτονται από τι κοινωνικέ δαπάνε, την παιδεία και την αγία. Πώ να μην διορωτούνται οι πολίτε τη Ένωση γιατί υπάρχουν 38,5 δισεκατομμύρια ευρώ για το νέο Ταμείο για την Άμυνα, ενώ κλείνουν τα γεροκομεία στη Φιλανδία. Η Ένωση χρειάζεται μια τολμηρή πολιτική για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Σήμερα η βιομηχανία καθορίζει τι πολιτικέ για το κλίμα σύμφωνα με τι δικέ τη ανάγκε. Οι λαοί όμω απαιτούν πραγματικέ λύσει. Απαιτούν πολιτικέ αποφάσει που να θέτουν φραγμό στην ανεξέλεκτη και ασίδωτη δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και δεσμευτικού στόχου για προστασία του περιβάλλοντο και αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή ακόμα πιο φιλόδοξου στόχου από τη συμφωνία του παρισιού. τέλο η ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική ασύλου και μετανάστευση βασισμένη στο διεθνέ δίκαιο στην ανθρωπιστική αλληλεγγύη προ του πρόσφυγε αλλά και την αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη. χρειάζεται να δημιουργεί ένα μόνιμο μηχανισμό για τη φιλοξενία όλων των προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη ανάλογα με τι δυνατότητε του καθενό κύριε πρωθυπουργέ για να γίνουν αυτά χρειαζόμαστε μια άλλη ευρώπη την ευρώπη για την οποία η αριστερά παλεύει την ευρώπη της ειρήνης της πραγματικής αλληλεγγύης της κοινωνικής δικαιοσύνης την ευρώπη των λαών. ευχαριστώ πρόεδρε. Ευρώπη για τη Δημοκρατία και την ε, Άμεση Δημοκρατία, η κυρία Νταμάτο, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περάσει από μια ριζική διαδικασία αλλαγής. Αυτή που απαιτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες όλο και πιο έντονα είναι παντού ορατά τα μηνύματα, οι δυνάμεις του κατεστημένου, τα κόμματα, τα φιλελεύθερα και τα σοσιαλιστικά χάνουν διαρκώς τις εκλογικές αναμετρήσεις. Οι πολίτες έχουν πλέον κουραστεί από την ε, αδικία, από τη ε, λιτότητα, από την διαφθορά και θέλουν την αλλαγή πλέον στις κυβερνήσεις των χωρών τους. Ε, έχουν στείλει λοιπόν πολλές φορές τους ε, προηγούμενους ηγέτες ε, στα σπίτια τους. Στην Ιταλία λοιπόν, η... για να σας δώσω μια εικόνα, η οικονομική πολιτική ήταν ισοδύναμη με μια οικονομική σφαγή, με μια καταστροφή. Όμως εμείς τώρα Κάνουμε προπολογισμό ο οποίος δίνει δύναμη στον πολίτη, ο οποίος δίνει νέες επενδύσεις, ο οποίος περιορίζει τις την διασπάθηση χρήματος. Έχουμε ένα επίδομα κατώτατο στήριξη των εισοδημάτων, το οποίο η Φινλανδία το γνωρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίς να θέλουμε να κάνουμε πολιτική πρόνοια, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την αγορά εργασίας, αλλά θέλουμε να μειώσουμε και τη φτώχεια. Πάνω από 5 εκατομμύρια είναι η φτωχοί στην ε, Ιταλία. Νέες δεξιότητες θα εξασφαλίσουμε για αυτούς που δεν έχουν θέση εργασίας και έτσι θα αυξήσουμε την απασχόληση με ένα πιο εξειδικευμένο ε, εργατικό δυναμικό που θα διευκολύνεται έτσι και η πρόσληψή του θα ενισχυθεί χάρη σε αυτή την ενίσχυση εισοδήματο ε, και εσωτερική κατανάλωση. Μια Ιταλία λοιπόν ενωμένη, μια Ευρώπη ενωμένη, αλλά και αλληλέγγυα. Ε, ήταν πολλοί οι ψευτοπροφήτες της αλλαγής, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτοί ε, οι οποίοι υποτάσσονταν στα λόμπι, όπως ο Μακρόν είναι παραδείγματι, όπως το θέμα της γλυφοζάτης στην Γεωργία, που δεν θα, το, δεν θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτό πριν από μερικά χρόνια. Δεν μπόρεσε να μας κοροϊδέψει ο Μακρόν. Ακολούθησε τις υποδείξεις της ε, ε, Μέρκελ και ενέκρινε την παράταση χρήσης του ισκληφοζάτης ε, για λογαριασμό της Bayer που εξεγόρασε τη Μονσάντο το 2018. Ας σταματήσει λοιπόν αυτή η υποκρισία, Ο πολιτή θέλει να δει πραγματικά και πράξεις, γεγονότα. Θέλει μια Ευρώπη που θα έχει παγκόσμια αντανάκλαση, θα μιλάει με μια ενωμένη φωνή, μια μόνη φωνή και βεβαίω χρειάζεται μια ε, έδρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλεία, αλλά η Μέρκελ και ο Μακρόν κάθονται χώρια και συζητούν μόνοι του για το μέλλον το οποίο θέλουν να χαράξουν οι δυο του ενώ θα το πληρώνουν οι 27. Και έτσι αποκλείουν τα 50 τα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Αλλά δεν μπορούν αυτοί οι δύο να φτιάξουν, έστω και αν φτιάξουν ενότητα άμυνας, ένωση άμυνας, την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται η συμμετοχή ολόκληρης της ε, Υπήρου. Η Ιταλία χωρίς να έχει ηγεμονικές διαθέσεις είναι η τρίτη μεγαλύτερη δύναμη, είναι όμως εγγυήτρια ε, στην Ευρώπη για την... Ε, ενότητα για την αλληλεγγύη και έτσι θέλουμε μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να περιλάβει και τις, ε, τα θεσμικά όργανα, χωρίς όμως παρεμβατισμό, χωρίς διευθυντική συμπεριφορά που θα εξασφαλίζουν την ενότητα που δεν θα κρατάνε τις Βεξέλλες μακριά από τον πολίτη γιατί αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όχι φτιάχνοντας ακόμα ένα χωριστό κύκλο λήψη αποφάσεων, αλλά επαναφέροντας την διαδικασία λήψη αποφάσεων στο μόνο άμεσα εκλεγμένο όργανο που εκπροσωπεί τον πολίτη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν θέλει να αλλάξει η Ευρώπη, πρέπει και να εγκαταλείψει τις πολιτικές λιτότητας που καταστρέφουν την εκπαίδευση, την υγεία, τη δημόσια, τα δικαιώματα και να σταματήσουν οι αυτοκριτικές, οι ψεύτικες του Γιουνκέρ για τα λάθη, γιατί οι δρόμοι που ακολουθείτε είναι πάντα οι ίδιοι και απευθύνω έκλεισε σας αγαπητοί συνάδελφοι, α κατασ... απορρίψουμε τη μακροοικονομική ε, προσέγγιση, την μακροπροληπτική προσέγγιση. Ας αφήσουμε κατά μέρος αυτές τις υποδείξεις των Βρυξελών, να προστατέψουμε περισσότερο τους πολίτες. Είναι απαραίτητο αυτό και για την ανάπτυξη των χωρών μας, των περιοχών μας, για την ε, αντιμετώπιση των προβλημάτων των περιβαλλοντικών. Πρέπει η Ευρώπη και μπορεί να αλλάξει αν είναι στο πλευρό του πολίτη και αν μπορεί να τους δίνει απαντήσεις και όχι προβλήματα συνέχεια και κολάφους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποργέτσιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε. Φαντάζομαι ότι σας ε, ξαφνιάζει λίγο αυτή η συμπάθεια που δείχνουν όλοι οι Ευρωπαίοι προς την ε, χώρα σας, όπως εκφράστηκε εδώ μέσα και ίσως πρέπει να κοιτάξουμε ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι, αυτούς που εσείς ονομάζετε λαϊκιστές, έχουν κάποιες επιφυλάξεις, γιατί όταν λέτε ότι είστε σε θέση να υποδεχθείτε 20-25 χιλιάδες πρόσφυγες, τη δική μας δουλειά κάνετε, γιατί βλέπουμε ότι ε, αυξάνεται η συνείδηση του πολίτη που δεν είναι ρατσιστής, που δεν είναι ξενόφοβος, αλλά που βλέπει ότι αυτή η άτακτη μετανάστευση αποτελεί ε, πηγή ανασφάλειας, δυσκολιών στην κοινωνική ένταξη, προβλημάτων τρομακτικών και ίσως θα ήταν πολύ πιο ευφυές και φρόνιμο να πει κανείς, όπως άλλωστε έχουν πει και κάποιοι από την ηγεσία του Κοινοβουλίου, θα ήταν καλό να προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο Μάρσαλ για την Αφρική. για τη σωστή λύση, η σωστή συνταγή δεν είναι η υποδοχή στις δικές μας χώρες και κοινωνίες με μια διαδικασία ένταξης που είναι πολύ αργή αλλά και αδύνατη μερικές φορές αν αναφερθούμε σε ορισμένους που προέρχονται από περιοχές και πολιτισμό μουσουλμανικό επί παραδείγματι που είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν στις κοινωνίες μας αλλά θα ήθελα ιδιαίτερος ε, για εσά που εκπροσωπείτε μια χώρα πλούσια και ένα μεγάλο λαό, ε, τη Φιλανδία, ε, να μας πείτε τι έχετε να πείτε για ένα σχέδιο Μάρσαλ που θα μπορούσε να εισαχθεί. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αυτή η Ευρώπη, η οποία έχει χάσει κάπως τον δρόμο της, είναι κάπως υποτίθεται ε, λαϊκιστική, ε, όπως λέγεται ε, δημαγωγική, που όμως αναζητεί ένα ρόλο ιστορικό που της ανήκει να βοηθήσει τους αφρικανικούς λαούς, όχι όπως το παρελθόν όμως, χρηματοδοτώντας πολέμους και κερδοσκοπία, αλλά με πραγματική γνήσια υποστήριξη, που ίσως να περάσει και από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτούς που, τους επιχειρηματίες που ξέρουν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους με σωστό τρόπο και που έτσι μπορούν να ξεριζώσουν και το πρόβλημα της μετανάστευσης και συγχωρέστε μου την έκφραση δημαγωγική ήταν η δική σας η προσέγγιση στην ε, μετανάστευση ήταν δημαγωγική όλη αυτή και αν εγώ ήμουν αγνήσιος πραγματικός ε, Φινλανδός θα είχα επιλέξει να αλλάξω δρόμο. Αυτό που έχουν κάνει κάποιοι άλλοι με θάρρος στην Ευρώπη που μπορεί να κατηγορηθούν για ανεξογονοφοβία και ρατσισμό αλλά στην πραγματικότητα να ζητούν το γνήσιο δρόμο, το στον πραγματικό δρόμο, το δρόμο των δικών μας ιεραποστόλων που πήγαν μέχρι την Αφρική για να τους προσφέρουν πολιτισμό και εκπαίδευση να τους δείξουν το δρόμο. Ο Ντόν Μπόσκο, ο ιερέας που αν ζούσε ακόμα σήμερα όπως έγινε στο 19ο αιώνα στην ε, Ιταλία θα είχε δείξει τον τρόπο να δουλεύουμε, να αρχίζουμε να κάνουμε επιχειρήσεις και όχι να ερχόμαστε, να έρχονται εδώ στη χώρα μας, στις χώρες μας, να κλέψουν και να βιάσουν γιατί ποτέ αυτοί οι άνθρωποι στην Αφρική δεν έμαθαν να δουλεύουν σωστά και αυτό είναι το το σφάλμα, η υπετιότητα των εγκλημάτων που διαπράττουν αυτοί οι μετανάστε είναι δική σα, εσεί, που ποτέ δεν δώσατε την εκπαίδευση αυτού του λαού, Ο κύριο Φοντούλη με εγγεγραμμένο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρωθυπουργέ, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Το κυριότερο όμω είναι η πατερναλιστική αντίληψη που τίνει να εδρεωθεί σε πολλέ από τι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στου ευρωπαϊκού θεσμού. Οι ηγέτε τη Ενώσεω λειτουργούν σαν να κατέχουν εκείνη την απόλυτη αλήθεια και προσπαθούν να επιβάλλουν την ιδεολογία του πολίτε πολλέ από τι αποφάσει των ηγετών είναι μη αναστρέψιμε δημιουργώντα στου πολίτε την αίσθηση πω ο δημοκρατικό έλεγχο μέσω των εκλογών είναι ανώφελο. χαρακτηριστικό και πολύ πρόσφατο παράδειγμα η συμφωνία των πρεσπών η οποία μάλιστα χαιρετίστηκε από το σύνολο των ευρωπαίων ηγετών. ο ελληνικό λαό εξέφρασε την ξεκάθαρη αντίθεσή του όμω η κυβέρνηση τσίπρα αδιαφόρησε δημιουργώντα τετελεσμένα. συντασσόμενη η ευρώπη πίσω από τη συμφωνία αυτή περιφρονεί τη βούληση των ελλήνων εμφανίζεται δέω εχθρική προ τα ελληνικά συμφέροντα θα ήθελα να υπενθυμίσω τόσο σε εσά όσο και στου υπόλοιπου ηγέτε τη Ενώσεω και ιδιαίτερο στον κύριο τσίπρα πως η εξουσία σας πηγάζει από το λαό και έχει ισχύ μόνο όσο ο λαός συνεχίζει να την εγκρίνει. σύντομα όμως θα διαπιστώσετε πως η εκ μέρου σα απαξίωση των ευρωπαϊκών εθνών θα αφυπνίσει τους πολίτες και θα του κάνει να σκεφτούν εθνικά. ευχαριστώ έχει το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα που το απευθύνθηκαν ο Πρωθυπουργό Φιλανδία. Παρακαλώ. Mr. President, thank you Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ομιλίες. Ε, θα απαντήσω στις ερωτήσεις σύντομα. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ Ζαν Κλόντ και Γιούρκη για τα καλά σας λόγια. Και Βεβαίω και εγώ να σου πω ήταν μεγάλη μου ευχαρίστηση η συνεργασία με την Κομισιόν. Η γεγονό είναι πως ε, θα είναι δύσκολη η στιγμή που θα αναλάβουμε την Προεδρία. Θα έχουμε μια Κομισιόν, ε, θα έχουν γίνει ευρωεκλογέ, θα έχουν γίνει και οι δικές μας εκλογές πριν. Πριν από αυτό θα έχουμε τις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ, το Brexit, ε, ο ΝΕ και τα λοιπά. Μεγάλα θέματα. Ζαν Κλοντ, ε, επίσης ε, είχατε δίκιο για τα ζητήματα της Αρκτικής ε, και την κλιματική αλλαγή. Εμείς είμαστε έτοιμοι για την Αρκτική Σύνοδο Κορυφής σε λίγες εβδομάδες. Το επενδυτικό ταμείο του Γιούρκη Κατάινεν είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο και στη Φιλανδία. Κύριε Βέμπερ, συγχαρητήρια για τον ε, ορισμό σας. Η συνεδρίαση του ΕΛΚ στο Ελσίνκι ήταν θετική και για εμένα, καθώς ε, συνάντησα γύρω στους 10 συναδέλφους ταυτόχρονα. Συμφωνώ μαζί σας για τις οικονομικές αρχές για ε, το ΠΔΠ το έχω ήδη συζητήσει με 17 συναδέλφους ε, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και οπωσδήποτε θα βρεθεί μια συμβαστική λύση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Για την κλιματική αλλαγή συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για να μπορεί ο κόσμος ε, να την δεχτεί και τονίζω ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να κάνουν περισσότερα από ό,τι νομίζαμε. Π.χ. υπάρχει η δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα, υπάρχει ένα μικρό πανεπιστήμιο εκεί στην ε, Λαπωνία, ε, πιάνουν το διοξίδιο του άνθρακα από τον αέρα και φτιάχνουν προϊόντα διάφορα. Και επίσης ε, και η χαμηλή τιμή της ηλιακής ενέργειας έχει μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε λοιπόν το τι δυνατότητες δίνει αυτό στην ε, Αφρική. Κύριε Κόφοντ, μάθετε φιλανδικά νομίζω στην ομάδα σας. Έχετε κάποιους φιλανδούς. Καλό είναι αυτό. η ευτυχέστερη χώρα στον κόσμο η Φιλανδία μπορεί να είναι αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι είμαστε και αυτοί που το κρύβουμε καλύτερα αν δείτε τις συζητήσεις στο εσωτερικό μας. Ανέφερα τον κοινωνικό πυλώνα. Επίσης, οι προτεραιότητες μας είναι η ισότητα των φίλων Έχουμε παίξει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτών με τον Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που δώσαν πολιτικά δικαιώματα στις ε, γυναίκες. Φορολογική παράδειση. Συμφωνώ πλήρω με αυτά τα οποία είπατε. Πρέπει αυτό να αφορά όλες τις εταιρείε και όλους τους ε, πολίτες, ε, δηλαδή να πληρώνουν όλοι φόρους εκεί όπου παράγονται τα κέρδη. Αυτή είναι μια βασική αρχή. Κύριε Ρούχονεν Λέρνερ, θα απαντήσω στα φιλανδικά, αν θέλετε. Και σε αυτό το φόρουμ ε, είναι καλό νομίζω να ε, επαναλάβω το τι εννοούσα όταν είπα ότι διαθέτω το σπίτι μου. Ξέρετε ότι ε, είχα μια οικογένεια την οποία φιλοξένησα πράγματι γιατί είχε κάποια συνεργασία με το εξωτερικό στη χώρα της και ήταν χριστιανή σε μουσουλμανική χώρα και κινδύνευε η ζωή τους ε, κάθε μέρα. Ε, δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς ζούσαν πριν φύγουν η οικογένεια αυτή ήθελε να ε, έρθει να εγκατασταθεί στο σπίτι μου και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάναμε στην Φινλανδία σε μια τέτοια ατμόσφαιρα όπου θα έπρεπε τελικά να ανακαλέσω αυτή την οικογένεια για να προστα... την απόφαση για να προστατεύσω την οικογένεια αυτή γιατί μου είπε η αστυνομία ότι δεν ήταν ασφαλής η οικογένεια αυτή στο σπίτι μου. Γι' αυτό τελικά αναγκάστηκαν να μετακομίσουν αλλού. Μετά, α, άλλος... έφυγε, έχει και δουλειές. Λοιπόν, να απαντήσω στην ε, κυρία Κέλλερ. Έχω εργαστεί και σε προσωπικό επίπεδο για τα ζητήματα κλιματικής ε, αλλαγής και έχω υποσχεθεί η οικογένειά μου θα είναι ουδέτερη ως προς το διοξείδιο του άνθρακα στο τέλος του επομένου έτους. Έχω ηλιακά πάνελ, έχω ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχω μειώσει την κατανάλωσή μου και έχω φυτέψει και τα σχετικά δέντρα. Οπότε το αποτέλεσμα τελικά είναι ουδέτερο. Αλλά είναι πολύ εύκολο για ένα άτομο να το κάνει. τότε χρειάζεται κοινή δράση σε τρεις τομείς, σε τρεις μορφές. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές και να συνεχίσουμε προς τα εκεί και βεβαίως να αυξηθούν οι καταβόθρες και ο φιναδικός τρόπος, ο βιώσιμος ε, διαχείρισης ε, του δάσους, είναι απόδειξη πως αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος ε, διαχείρισης και, αυτό είναι κάτι το οποίο στηρίζω. Επίσης ε, χαίρομαι για το ότι υπάρχουν νέοι τρόποι δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα από τον αέρα και αποτελεί πλέον πηγή άλλων προϊόντων. Και πρέπει βεβαίω να φυτεύουμε και δέντρα. Αναφέρατε ότι έχουμε κάποια εμπειρία συνεργασίας με λαϊκιστικά κόμματα. Ε, το μήνυμά μου είναι ότι και τα λαϊκιστικά κόμματα πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνες ε, κυβερνητικές. Και έτσι ε, έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Να αναλαμβάνουμε ευθύνες και έτσι θα απαντήσουμε, θα δώσουμε και απαντήσεις στον κόσμο. Αναφέρατε κύριε Σιλικιώτη. Το ότι ο Ιαλα, γνωστός φιλανδός αριστερός, είπε στην κοινοβουλία μας πως ο καλύτερος φίλος των φτωχών είναι ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Έτσι θα φροντίσουμε τους πάντες σε κάθε χώρα, κάθε μέρα. Γι' αυτό στην Φιλανδία τα επιδόματα είναι τόσο υψηλά πέρα από την ε, εκπαίδευση βεβαίω που είναι ίδια για όλους τους πολίτες μας. Κυρία Ανταμάτο, το ποσοστό απασχόλησης συμφωνώ ότι είναι βασικό για να ισορροπήσει η οικονομία και βεβαίως στηρίζω όλες τις ε, δράσεις ε, που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι εξαντλήθηκε ο χρόνος. Με ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία Κατσιάη. Πρώτος ομιλητής, μάλλον ομιλήτρια, είναι η κυρία Γιασλοβιάσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Πρωθυπουργέ, ε, θέλω να σας πω ότι η Προεδρία σας ε, είναι πολύ, ήταν πολύ ισόρροπη, μιλάτε πολύ για προστασία του περιβάλλοντος ε, και των πολιτών. Είστε Πρωθυπουργό σε μια χώρα η οποία έχει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη, για να μην πω παγκοσμίω. Ε, νόμιζα ότι θα μιλούσατε πολύ για εκπαίδευση, παρόλο που είναι ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν θα προτείνατε να επιβληθεί παντού το ε, φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα που προετοιμάζει σήμερα καλύτερα τους μαθητές και τους μελλοντικούς πολίτες. Ε, το κοινωνικό κεφάλαιο είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο ακόμα και στην οικονομία. Σήμερα έχουμε ρομποτοποίηση, αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη δεν θα πρέπει να προετοιμάσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν ε, ε, θα είναι προτεραιότητα αυτή της Φιλανδικής Προεδρίας. κυρία Καμπούλα Νάτρη. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητέ Πρωθυπουργέ, καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω ότι δεσμεύεται τόσο πολύ η μελλοντική Προεδρία προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, βλέπουμε παγκόσμιες προκλήσεις και μόνο ε, από κοινού μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Βλέπουν ότι από την άλλη πλευρά της μάχης προσπαθούν να πάρουν το δικό τους δρόμο, αλλά είναι πολλά τα προβλήματα ε, για να βρουν αυτό το δρόμο του Brexit στην πορεία τους. Επίσης, μας είπατε, κύριε Πρόεδρε, ότι ε, δεν είμαστε ε, προετοιμασμένοι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Είναι κοινή η στόχη, είναι κοινά τα προβλήματα και ο κόσμος περιμένει από εμάς να είμαστε πρωτοπόροι στην προσπάθεια αυτή. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στη νέα οικονομία. ο κύριος ε, Γιούγκερ ε, έχει αναφερθεί και ο ίδιος στη σημασία της Αρκτικής και της Βόρειας Ευρώπη. Δεν έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας μόνο προς Ανατολάς και προς Νότον, αλλά και προς την Αρκτική. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και ένα... Πρωθυπουργέ της ε, Φιλανδίας, κύριε Σίπηλα. Ήθελα να σας θέσω το θέμα της κοινή αμυντικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης. ξέρετε χθες είχαμε την θλιβερή επέτειο των ημείων. τα Ιμία είναι μια περιοχή που ανήκουν στην ελλάδα δύο νησιά που ανήκουν στην πατρίδα μου και όμως υπάρχουν οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις της τουρκίας. μάλιστα αυτές τις ημέρες τουρκικά πολεμικά περιπολούν στην περιοχή. η τουρκία συνεχίζει τις παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο στα ελληνικά χωρικά ύδατα απειλεί την ελλάδα με κάζους μπέλι σε περίπτωση που η ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Ο Ερντογάν θέλει να ανατρέψει τη συνθήκη της Λοζάνης και θέλω μια δήλωση σαφέστατη. Πρώτον, στήριξη της Ελλάδος απέναντι στις απειλές του Ερντογάν και της Τουρκίας. Και δεύτερον, τη θέση σας για να υπάρξει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίζει την Ελλάδα σε περίπτωση αμφισβήτησης των συνόρων της από την πλευρά της τουρκίας να υπάρξει στήριξη της ευρωπαϊκής ένωσης στα σύνορα της ελλάδος τα οποία είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και θέλουμε μια σαφέστατη τοποθέτηση από εσά κύριε πρωθυπουργέ εδώ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο γιατί θα είναι μήνυμα απέναντι στον ερντογκάν απέναντι στις απειλές της τουρκίας. σας ευχαριστώ. Grazie, Presidente. Κυρία Κατάινεν. Ναι, το έχω ανοίξει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Σίπηλα, ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που στην ομιλία, της, η ομιλία σας μιλήσατε για τον πραγματισμό που χρειάζεται, για τον ρεαλισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δράσεις της. Η ακαιρεότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οικονομική της βιωσιμότητα δέχεται πιέσεις από πολλές διαφορετικές πλευρές και υπάρχουν, ε, υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη να ξαναδούν σε νέα βάση τις μορφές συνεργασίας τους. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στο διεθνές προσκήνιο. Κύριε Πρωθυπουργέ, πώς νομίζετε ότι μπορεί να προωθηθεί η ιδέα, ας πούμε, ότι η οι κλιματικέ αλλαγέ και η κατανομή του βάρου του μεταναστευτικού φαινομένου θα πρέπει να γίνει πιο εξισορροπημένα μεταξύ των κρατών μελών. Διότι εγώ η ίδια βλέπω ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί μα. Και αυτό φαίνεται και από το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τι επερχόμενε ε, ευρωεκλογέ. Και ελπίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, στην ομιλία σας να διορθώσετε κάποιος παρανοήσεις για την ε, φιλανδική δασοκομεία και το κατά πόσο μπορεί να είναι βιώσιμο και στο μέλλον. Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο σε όλους όσοι ζήτησαν να παρέμβουν. Ωστόσο, θα πρέπει να σεβαστείτε το ένα λεπτό ομιλίας που έχει αποδοθεί στον καθένα σας. Ιδάλλως θα είμαι υποχρεωμένος να διακόπτω τις παρεμβάσεις γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίες. Ο κύριος Μπούκνερ. Κύριος Μπούκνερ, ευχαριστώ. Ε, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ και ένα χρόνο και πάνω από ένα χρόνο η κυβέρνησή σας μαζί με τη Γαλλία και 8 ακόμα χώρες μπλοκάρεται οποιαδήποτε πρόοδο στην καταπολέμηση εξαγωγής τεχνολογίας παρακολούθησης σε δικτατορίες. Πέρσι, η δική σας κυβέρνηση μαζί με άλλες πήρατε θέση κατά της προστασίας ε, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε είδη διτής χρήση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς το υπερψηφίσαμε με 92% πλειοψηφία και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέραμε μια πρόταση για να προστατέψουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είστε η επόμενη Προεδρία. Μέχρι σήμερα το Συμβούλιο έχει δράσει τελείως ανεύθυνα. Παγκοσμίως δημοσιογράφοι, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρακολουθούνται και ε, συλλαμβάνονται, φυλάσσονται και θανατώνονται με δική μας τεχνολογία. Ελπίζω να πάρετε σοβαρά ε, τις ευθύνες σας και να το αλλάξετε αυτό. Η κυρία Κίλλονεν Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί Ευρωπαίοι αισθάνονται ξένοι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να λοιπόν, γιατί οι λαϊκιστές βρίσκουν γόνιμο έδαφος. Όχι. Θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα πιο ανθρώπινα. Είτε μιλούμε για την απασχόληση, είτε για το κλίμα. Όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν, να δουν τι δυνατότητέ τους, να μην αισθάνονται ξένοι. Τι μπορεί να κάνει η χώρα σας ούτως ώστε να υπάρξει περισσότερη ισότητα, δικαιοσύνη, ε, κοινωνική ένταξη. Όχι μπορεί δηλαδή να ενστερνίζεται το, το θέμα ότι είναι, ότι είναι δική του η Ευρώπη. έχουμε μόνο την Ευρώπη τη οικονομίας και του χρήματος. Πρόεδρος κονσάρι. Arvoisa puhemies, κυριε Κύριε Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα καλώς ορίσατε Πρωθυπουργέ Σίπηλα ή στο Κοινοβούλιο. Μα ονομάζουν τη συνείδηση τη Ευρώπη γιατί ασχολούμεθα με ανθρώπινα δικαιώματα που τη σήμερα ημέρα είναι πολύ σημαντικό. Λίγο με απογοητεύσατε από όσα είπατε πάντω όσον αφορά τα οικονομικά. Τι γίνεται όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία μια η φιλανδία και πάλι έχει τοποθετηθεί εν μέσω των ε, νεοφιλελευθέρων. Και τι γίνεται και για την μετανάστευση. Μας λέτε για επαναπατρισμούς. Κάπου κάπως αλλάξατε νομίζω τον τόνο, αλλάξατε την κατεύθυνση των εξαγγελιών σας. θα πρέπει να συζητούμε όλα τα θέματα και όχι μόνο το πώ θα καταστεί δυνατόν να στείλουμε πίσω αυτού του ανθρώπους στην ε, χώρα τους. Πάντως, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την Κομισιόν και το Συμβούλιο που είπατε τα θέματα της Αρκτικής, γιατί και στην Αρκτική η συνεργασία με την Ρωσία πάει καλά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, λόγω στον ε, επόμενο. Ευχαριστώ, έχω δύο θέματα να έχω δύο προτάσεις προς τον Φιλανδό Πρόεδρο και τον ευχαριστώ πρώτα πρώτα την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης σχετικά δηλαδή με αυτό το οποίο συμβαίνει σαν ένα σπουδαίο λαό, σε τον μεγάλο λαό της Βενεζουέλας όλα αυτά τα οποία τώρα υποφέρουν σχετικά με αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να δείξουμε ότι ασπαζόμαστε δημοκρατία ε, η ειρήνη ούτως ώστε να υπάρχει ελευθερία, πολιτικά δικαιώματα για όλους, να προστατεύονται γυναίκες, ανήλικοι. Ε, εσείς τι πιστεύετε σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να αναγνωρίσετε τον ε, νέο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά τον και όσον αφορά τον αθέμητο ανταγωνισμό, την οικονομία και το διεθνές εμπόριο. Κατέστη δυνατόν να αποσπάσουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα ε, και να μην χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας περισσότερη πλαισίωση. Ιωάννα. Micro, please. Micro. Το μικρόφωνο σας λέει ο πρόεδρος. Domnule prim-ministru, mă bucur că ne aflăm astăzi aici. Χαίρομαι, κύριε Πρωθυπουργέ, που σήμερα συζητούμε ζήσα εσεί ω Φιλανδό Πρωθυπουργό και εγώ ως Ευρωβουλευτή εκπροσωπώντα την χώρα που τώρα ασκεί την ε, Προεδρία του Συμβουλίου της ε, Ένωσης. Όλα αυτά σα τα λέω γιατί πρόκειψαν διάφορα σκάνδαλα. Σκάνδαλα για κάποιε δηλώσει που λέγατε ότι είσαστε έτοιμοι να λάβετε την Προεδρία κατευθείαν από τη Βουλγαρία και έτσι να βάλετε σε παρένθεση τη δική μα. Ναι, βεβαίω. Είδατε τις δηλώσεις μας ε, και είδατε ότι μόνο η κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει την ε, Προεδρία. Δηλαδή θα πρέπει να λάβετε υπόψη μόνο τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και όχι άλλες δηλώσεις. Είμαι πεπισμένος ότι τώρα που παρήλθαν κάποιοι μήνες μετά από αυτές τις απρεπείς δηλώσεις ότι έχετε αλλάξει ρότα και έναν μήνα μετά την άλεψη της Προεδρίας η χώρα μας ήδη έχει κλείσει διάφορα σημαντικά ζητήματα. Το μήνυμά μου είναι η συνέχεια. Ελπίζω να συνεχίσετε το έργο της Ρουμανικής Προεδρίας. Επόμενος. Ευχαριστώ και συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προαγάγει μέσω της εξωτερική πολιτική διάφορε αξίε, να προστατεύονται αυτές τις αξίες όμως και στο εσωτερικό τη χώρα. Δεν θα πρέπει αυτές οι αξίες να ερμηνεύονται αυθαίρετα, ούτε θα πρέπει ε, οι Βρυξέλλες να ε, υπαγορεύουν πώς θα υλοποιούνται αυτές οι κοινέ αξίες αυτές που ενώνουν όλο τον κόσμο. Τώρα όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς, πιέζεται κάποια κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ε, ε, κάποια μοντέλα φιλελεύθερα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μας ενώνουν. Ε, θα πρέπει να φέρουν φέρνουν πιο κοντά. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ο μπαμπούλα Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία, αλλά ενωμένοι δεν είμαστε στην πραγματικότητα είμαστε διαφορετικοί και αυτό θα πρέπει να το αποδεχθούμε και θα πρέπει επομένως να βαδίσουμε με πηξίδα την επικουρικότητα. Ο επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στο κοινοβούλιο κύριε Πρωθυπουργέ. Συνήθως λέμε ότι είναι απλό Ε, να βλέπει κανείς το τι δεν πάει καλά στον απέναντί του. Ε, αλλά εδώ μιλήσατε για ισοσκελισμένο προπολογισμό και μιλήσατε και τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ε, μαθηματική προσέγγιση που θα έπρεπε να έχουμε στην καθημερινή διοργάνωσή μας. Η Φινλανδία θα πρέπει να βοηθήσει και την Προεδρία που έχει αναλάβει να προωθήσει το ναι. θέμα αυτό και θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τη Φινλανδία στην Προεδρία της. Ευχαριστώ κυρία Χάουταλα. Kiitos puhemies ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Πρωθυπουργέ. Ο κύριος Πρόεδρος έχει πει ότι ακόμη και κάποιε από τι ιδρυτικέ ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να μάθουν ε, πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι χτίζεται στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θέλω να ρωτήσω δύο διαφορετικά πράγματα. Ποια είναι η φιλανδική στάση και τι δυνατότητε υπάρχουν για το πώς ε, θα εξετάζονται οι φορολογικές συμφωνίες μεταξύ χωρών. Ε, κάποιες χώρες δεν μπορούν να λάβουν μέτρα εναντίον άλλων που αποφασίζουν διμερώς να ε, έρθουν σε φορολογικές συμφωνίες. Όμως πρέπει να πατάξουμε και τη φοροδιαφυγή. Ξέρω ότι το συζητάτε το θέμα στο Συμβούλιο, όμως η Φιλανδία δεν φαίνεται να υποστηρίζει την κίνηση αυτή, διότι αντίκειται στην εθνική κυριαρχία των κρατών Και μετά υπάρχει και το θέμα τη εταιρική ευθύνη στην Φιλανδία. Είμαστε πολύ ενεργοί στο να υπάρχει μια νομοθεσία για τα θέματα τη εταιρική ευθύνη. Οι εταιρείε θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσει για τι συνέπειε των δραστηριότητών του στο περιβάλλον και σε άλλα θέματα. Και είναι σημαντικό αυτό για να τεθεί ω προτεραιότητα στη Φιλανδική Προεδρία. Ευχαριστώ. Κύριε Κούναν, ευχαριστώ Πρόεδρε, Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα ε, τη χρονιά που προετοιμάζεται για την τρίτη της Προεδρία η Φιλανδία και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις φιλανδικές προτεραιότητες. Πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει ενώ και απογοητεύτηκα λίγο. Γιατί δεν μιλήσατε πολύ για την έρευνα και για την εκπαίδευση, για την παιδεία. Το success story της Φιλανδίας ακριβώς εκεί βασίζεται, στο πάρα πολύ καλό εκπαιδευτικό μας σύστημα, το know-how, την τεχνογνωσία και την επένδυση στην καινοτομία που μας έχει κάνει από τις πιο καινοτόμες χώρες. Αυτά ακριβώς χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη, ε, ε, ανταγωνιστικότητα σε μια ψηφιακή οικονομία που αλλάζει τον κόσμο. Ε, ρομποτοποίηση, αυτοματοποίηση, αλλάζει ακόμα και η αγορά εργασίας. Εκεί είναι οι μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες προκλήσεις και γι' αυτό ε, αναφερθήκατε και στην κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση της. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ ε, εστίαση στην παιδεία, στην τεχνογνωσία, στην ποιοτική έρευνα και αυτό είναι το μήνυμά μας και για την επόμενη Προεδρία. Ήθελε το Κοινοβούλιο να αυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα η Φιλανδία έχει αυξήσει τις δικές της δαπάνες, αλλά τι γίνεται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συμφωνήσετε με την πρόταση του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις αυτές. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σήμερα συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης και νομίζω ότι έχουμε δύο επαναστάσεις οι οποίες πρόκειται να σημαδεύσουν τη ζωή μας σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης. Η τεχνολογική, η ψηφιακή και η ενεργειακή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και όσον αφορά την ενεργειακή επανάσταση που θα μας ε, σημαδέψει είναι ένα ορόσημο για το, το, τα ταξίδια, για την κατανάλωση θα πρέπει να δειχθούμε ε, φιλόδοξη επίσης για την αλλαγή του κλίματος. Κατά αυτή την ε, θητεία έγιναν πολύ σημαντικά βήματα και έτσι η Ευρώπη να γίνει πρωτοπόρα σε αυτή την ε, ενεργειακή μετάβαση, ούτως ώστε να απαλλαγούμε από τον ε, άνθρακα και να πετύχουμε τους στόχους για το κλίμα. Δεν θα πρέπει όμως να καταθέσουν τα όπλα ή να χαλαρώσουμε γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα και θα πρέπει η ανταπόκρισή μας να είναι συνεχής. Κατσέρσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει οικοδομηθεί. Και διαρκώς υπονομεύεται. Ε, υπάρχουν όμως και άλλες ε, θεμέλιες λύθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ενιαία αγορά, η αγορά εμπορευμάτων και ε, προσφοράς υπηρεσιών. είναι σαφές ότι κάποιοι θέλουν να παραβιάσουν την ελεύθερη κυκλοφορία. και όμως Είναι σημαντική η ελευθερία κυκλοφορία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται πέντε μέρε ε, για να πάει ένα φορτηγό από τη Φινλανδία στην επικράτεια τη υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Φινλανδοί ευρωβουλευτέ ήδη ε, πλήρωσαν για να μην χρησιμοποιηθούν να κατεξοδούν τι πράξει στο πακέτο τη ε, κινητικότητα. Εσείς μπορείτε να υποστηρίξετε τη λύση του Συμβουλίου. Δεν θα περιορίζατε έτσι τις ελευθερίες των πολιτών, τις οικονομικές τους ελευθερίες. Δεν θα άρετε έτσι οικονομικούς φραγμούς, ενώ έχουμε πει πανελειμμένως ότι οι φραγμοί αυτοί πρέπει να έρθουν. Είναι πολλές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να κλείσουν, να κατεβάσουν ρολά, οι Φιλανδοί καταναλωτέ θα πληρώσουν το τηλεπιτερή ε, για τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε κυρία Γκραπίνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρωθυπουργέ, ε, συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε ε, την συνοχή της ε, ενιαίας αγοράς, το κράτος δικαίου. Ήθελα εδώ όμω να θυμίσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν τη χώρα σας. Είπατε ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να υπάρξουν ε, νέα σύμφωνα για το κράτος δικαίου. Όμως στην χώρα σας δεν εφαρμόζεται πλήρως το κράτος δικαίου. Ξέρετε ότι βάσει της φιλανδικής νομοθεσίας έχουν, ε, υπάρχουν οικογένειες που τους έχουν πάρει τα παιδιά έχουν ε, προσφύγει στα δικαστήρια και δεν μπορούν να παρουσιαστούν ε, στην εκδίκαση της υπόθεσής τους. Εγώ κατα... έχω συντάξει σχετική υποστολή. Ε, τι μπορεί να γίνει όταν τέτοιοι Ευρωπαίοι πολίτες με ευρωπαϊκή θα γίνει άλλη της χώρας σας δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των Φιλανδών πολιτών. Θέλουμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση στο θέμα αυτό. Και επίσης, τι προϋποθέσεις μπορείτε να δημιουργήσετε για το κράτο δικαίου στη χώρα σας, γιατί βλέπω ότι ανάλογα με τη χώρα ε, το προσδιορίζετε διαφορετικά. Ευχαριστούμε. Ε, ε, κύριε Πρωθυπουργέ, η ομιλία σας ήταν ε, πολύ πραγματιστική. Ε, βασίζεται σε πολύ καλά στοιχεία και δίνει και μια πρόπτικη για το μέλλον. Μιλήσατε για τη δασοκομεία και τι προοπτικέ τη. Περίπου το 70% τη Φιλανδία καλύπτεται από δάση. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερε γνώσει στον τομέα αυτό. Και ξέρουμε και πώ να διαχειριστούμε με βιώσιμο τρόπο τα δάση. Τα δάση είναι πόρο για την Ευρώπη και την Αφρική. Ε, είναι πνεύμονας και επίσης ε, προσφέρουν θέσεις απασχόλησης και πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές. Σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο όμως θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και προς την Αρκτική και τα θέματα της Σκανδιναβίας γενικότερα. Στην περιοχή της Αρκτικής όπου ζω εγώ ίδια υπάρχει τεράστιο δυναμικό και φοβερή φυσική πόρη, ε, τρομερή τεχνογνωσία επίσης, αλλά και εδώ Πρέπει να αξιοποιήσουμε τους πόρους. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση στα θέματα της Αρκτικής. Ευχαριστούμε, ο κύριος Πόλτσακ. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ, Πρωθυπουργέ Σιπίλα, που ήρθατε για να μας δείξετε ότι η Φιλανδία είναι μια ευτυχισμένη χώρα μετά από 25 χρόνια συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το 1% του πληθυσμού. Θέλω να μιλήσω για τον Πολ Αρή Σπακ που είπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά κράτη. Όλοι μικροί είμαστε για τις προκλήσεις. Απλώς μερικές χώρε ξέρουν ότι είναι μικρέ και κάποιες άλλες δεν το γνωρίζουν ακόμα. Αυτά έλεγε ο τότε Βέλγος Πρωθυπουργό από τους πατέρες ιδρυτές. Μιλήσατε για τις, ε, την πολιτική άμυνα που είναι πρόκληση για σας και πρόβλημα που είστε ουδέτερη χώρα, αλλά δεν μιλήσατε για τη μετανάστευση. Παρακαλώ ενώστε τις δυνάμεις σας για να απεμπλακεί ο κανονισμός του Δουβλίνου όπως ήταν εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται κοινή πολιτική, χρειάζεται αλληλεγγύη για τη μετανάστευση. Καμία χώρα δεν μπορεί να τυφλή και να γεννάει από την άλλη όταν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη μας χτυπούν την πόρτα. Η κυρία Γιατενμάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ Σίπηλα θα διαπιστώσατε ότι είστε πάρα πολύ ευπρόσδεκτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί οι βουλευτές έχουν τόσες πολλές ερωτήσεις και οι Φιλανδοί οι ίδιοι βουλευτές που ε, νομίζουμε ότι είμαστε στη Φιλανδική ε, Βουλή στην ώρα των ερωτήσεων του Πρωθυπουργού. Ε, εμείς είμαστε εδώ ίσως πιο ευπρεπείς από τους Φιλανδούς συναδέλφους, δεν φωνασκούμε. αλλά τι γίνεται με την υλοποίηση και την εφαρμογή των αποφάσεων. Συμφωνώ μαζί σας, το είπατε κι εσείς. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάνουμε βήματα, παίρνουμε φιλόδοξες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ακολουθούν στη συνέχεια τα κράτη-μέλη ε, με την εφαρμογή τους. Τι θα πρέπει να γίνει. Πρέπει να αλλάξουν τακτική τα κράτη-μέλη. Πρέπει όλοι να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των νομοθεσιών. Οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι αρκετά καλά προετοιμασμένες ε, στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ε, εκεί που συνεδριάζουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων γιατί είναι αρκετά περίεργο αυτό. Μετά από τα συμβούλια ε, βγαίνουν διάφορες δηλώσεις, τι σπουδαία ήταν η συνεργασία και τι καλά που τα συμφωνήσαμε και μετά γυρνάνε στις πρωτεύουσε τους και δεν δίνουν συνέχεια. Θα φροντίσετε αυτές οι κενές αποφάσεις να εφαρμόζονται. Κάντε ησυχία σας παρακαλώ ο Πρόεδρος στα αγγλικά και καθίστε κάτω. down, Now, the speech, the conclusion. Και τώρα θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της Φιλανδίας να κλείσει τη συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Σίπηλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Είμαστε συνηθισμένοι σε υποβολή ερωτήσεων. Κάθε πέμπτη το κάνουμε αυτό στο κοινοβούλιο μας. Όλοι οι υπουργοί οφείλουν να είναι παρόντες. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Αλλά μετά τις ερωτήσεις ακολουθούν οι απαντήσεις και θα πρέπει να ομαδοποιήσω τις ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα για την παιδεία. Η ισότητα στην παιδεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και το δημόσιο σχολείο είναι το καλύτερο και για πλούσιους και για φτωχούς. Όλοι οι Φιλανδοί, όλα τα παιδιά όλων των Φιλανδών πάνε στα ίδια σχολεία. Έχουμε τους καλύτερους δάσκαλους στον κόσμο και θα πρέπει ένα εκατομμύριο Φιλανδών να περάσουν από το σχολείο τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτή η πρόκληση νομίζω ισχύει για όλες τις χώρες της ε, Ένωσης. Είναι θέμα τεχνητής νοημοσύνης, είναι θέμα των αλλαγών Τώρα για την αλλαγή του κλίματος. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, για το ότι συμφωνήσατε με αυτά που είπα και για όσα έθιξα ένα από σένα στην ομιλία. Είναι πολύ σημαντική η υπόθεση αυτή για μας και ειδικότερα ανησυχούμε το ε, διοξείδιο του άνθρακος και ε, ε, αυτό είναι με διαπραγμάτευση με είπα και με Ρωσία. Οι χώρε αυτέ ενδιαφέρονται κάτι να κάνουν και αυτές για το κλίμα τώρα για τις επενδύσεις πρέπει να γίνουν σωστά Τώρα, όσον αφορά την ε, συνεργασία στην άμυνα, ή τι συνεργασίες αυτή εξ αρχή εμεί ε, θεωρούσαμε ότι είναι καλή ιδέα και θεωρούμε θετικό το ότι υπάρχει πρόοδο σε αυτό το μέτωπο. Τώρα, για την Τουρκία, περίπλοκα τα πράγματα είναι χώρα του ΝΑΤΟ, και είναι και θέμα το κράτος δικαίου στην χώρα που μας ανησυχεί έτσι όπως είναι η κατάσταση και βέβαια και το τι θα γίνει σε σχέση με την Κύπρο για την Ρωμανία. Ανέκαθεν ήμουν βέβαιος ότι η Ρωμανία θα τα πάει άριστα ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδατε αποδείξεις αυτών που σας λέω. Θέλουμε να υπάρχει δημοκρατία, εκλογές, ε, ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα και βέβαια η χώρα μας θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις και φυσικά θα κάνει για θα συμμορφωθεί με ό,τι αποφασίσει η Ένωση. Είχαμε πάρα πολλά τα οποία ρώτησαν οι συμπατριώτες μου, οπότε στα φιλανδικά θα σας πω τα υπόλοιπα. Ε, <clears throat> Πρώτα-πρώτα όσον αφορά τη βιώσιμη δασοκομεία. 70% ε, με 80% στη χώρα μας από τα δάση τα χρησιμοποιούμε και τέλος πάντων ε, φυτεύουμε περισσότερα από όσα κόβουμε. Πώς να είμαστε ε, αποτελεσματικοί και βέβαια την κατασκευή των προϊόντων από ξύλο, θα να τι θα γίνει με τη χρήση του άνθρακα. Τώρα για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με πολλές ερωτήσεις και ως επόμενη ή, επόμενη προεδρία επί τη βάση των όσων έχω πει με τους συναδέλφους θα μπορέσουμε να κλείσουμε έναν συμβιβασμό για τις παραδοσιακές κοινωτικές πολιτικές και για τις νέες προκλήσεις. επιδεικνύουμε ευελιξία στην πολιτική μας και ως Προεδρία νομίζω θα βρούμε τις πιο αυτοχές λύσεις όταν έρθει η ώρα. Για υλοποίηση, ε, τα είπα στην αρχή στην ε, εισήγησή μου και η παράδοσή μας είναι ότι όταν συμφωνούμε για κάποιο ζήτημα, ε, τότε τηρούμε τα υπεσχημένα. από την αρχή. Ε, νομίζω και για αυτό υπάρχουν αποδείξεις. Όταν αποφασίσουμε το κάνουμε με οριμότητα και στη συνέχεια προχωρούμε στην υλοποίηση της απόφασης. Ε, αυτό είναι το πιο ζουμερό μήνυμα της ε, ομιλίας μου. Ε, ευχαριστώ πρώτα, μεγάλη μου ευχαρίστηση να παραστώ σε αυτή την συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πάλι ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Prime Minister, thank you for your answer. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ για την απάντησή σας και για τη θέση σας ε, ε, για τη Βενεζουέλα. Η συζήτηση έχει λήξει. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες.